propose de reprendre euh, les débats pour, pas ne, pour ne pas prendre de retard sur... Να συνεχίσουμε τη συζήτηση για να μην καθυστερούμε. Ήδη έχουμε μείνει πίσω σχετικά με την ημέρα διάταξη πρώτα-πρώτα. Ε, η κυρία Σπέρ, με συγχωρείτε. Έπρεπε να λάβει το λόγο το πρωί, αλλά είχατε, δεν μπορούσατε να λάβετε το λόγο και τώρα είχατε καλοσύνη να κάτσετε να μας μιλήσετε τώρα για το απόγευμα. Είναι καθηγήτρια όσον αφορά τον σημερινό αραβικό κόσμο στο ελεύθερο μεσήμα των Βρυξελών και θα μας πει τι γίνεται στο Λίβανο σήμερα στον αφορά τον σχηματισμό κυβέρνησης. Όχι, δεν έχουμε χρόνο για ανταλλαγή απόψεων. Την άλλη μεριά. Απουσιάζει η αντιπροσωπεία του Λιβάνου. Επομένω, δεν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων αφού οι Λιβανέζοι φίλοι απουσιάζουν. Κύριε Σφέρ, έχετε το λόγο. Κάντε μας μια παρουσία σε σχέση με το τι γίνεται σήμερα στον Λίβανο. On m'a demandé de faire 10 minutes de présentation, donc je reviens de Beyrouth. παρουσίαση είπατε να κάνω. Λοιπόν, γύρω τώρα από την, ε, ε, από την Βίρτο, όπως γνωρίζετε όλοι στον Λίβανο, σήμερα έχουμε τη δεύτερη υπουργική κρίση. Όχι, δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη και ήδη έχουμε ένα πεντάμινο κατά το οποίο η, η κυβέρνηση ε, μόλις κατάφερε να σχηματίσει μια ε, κυβέρνηση και είναι τέτοια η κατάσταση που αντικατοπτρίζει την ε, συγκυρία αυτού του πολιτικού αδιεξόδου. Πρόκειται για μια σύγκρουση που ξεκινά από το 2005, οπότε ο πολιτικός κόσμος διχάστηκε και γνωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Πρώτα-πρώτα έχουμε το συνασπισμό, ας πούμε, της 14ης Μαρτίου και έχουμε επίσης τους ε, άλλους, ε, τους, τους ε, χριστιανούς και έχουμε επίσης και το άλλο στο του Χεσμολάχ και τους συμμάχους της. Το ΣΕΠΕΛ του στρατηγού Σελάν. Πρόκειται επομένως για κάποια εσωτερική πολιτική κρίση που σοβεί στο Λίβανο που επίσης αντικατοπτρίζει αυτό το, το, το, την ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Γνωρίζετε ότι το 2006 επετέθη το Ισραήλ στον Λίβανο, το 2008 τον Μάιο, κατόπιν επίσης ε, ε, μιας ε, κρίσης υπήρξαν μάχες, υπήρξε μάχη αντιπαραθέσεις στην, στην Βηρητό και ο Μισελ Λεμάν, ο επικεφαλής του στρατού είναι το σύμβολο της Εθνικής Ενότητας σήμερα. Οπότε θα έπρεπε να βρεθούν 30 άτομα να εξηγήσουν την κυβέρνηση, 15 για την πλειοψηφία, δηλαδή για το συνασπισμό της 14ης Μαρτίου και 10 για την μειονότητα, δηλαδή για την αντιπολίτευση, Χεσμολά, Χαμά και ΣΕΠΕΛ Και υπάρχουν και κάποια άλλα κόμματα τα οποία δεν τα ξέρω, τα, τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα. Και επίση άλλοι πέντε υπουργοί ε, πρόκειτο να αναλάβουν θόκου για τον πρόεδρο τη κυβέρνηση. Ο Τζουμπλάτ, ο επικεφαλή του Πρωθυπουργού Σοσιαλιστικού Κόμματο και πρόεδρο του συνασπισμού 14 ε, Μαρτίου, τώρα τελευταία προσέγγιζε την ε, Συρία και αποστασιοποιήθηκε από τον συνασπισμό και κατευθύνεται προς σχηματισμό ενός ρεύματος ε, κεντρώου. Αλλά σήμερα τα πράγματα έχουν διαφορετικά. Δεν έχουν πια τους 15 υπουργούς της πλειοψηφία, αλλά μάλλον έχουμε 12 συν 3. Τρει για τον Τζουμπλάτ, για, για, για, την κεντρώα παράταξη και άλλου 10 για την μειοψηφία, την αντιπολίτευση και, και άλλους ε, τους υπόλοιπους από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτές, αυτοί οι δύο συνασπισμοί αντιπροσωπεύουν διάφορες κοινότητες της ε, χώρας ε, και έχουν επικεφαλής κάποιον, κάποιον ηγεμόνα και γύρω γύρω υπάρχει ένα, ένα σύστημα πελατειακό σήμερα. Επομένως έχουμε τις διαπραγματεύσεις για τα χαρτοφυλάκια των Υπουργών για να δούμε τι αντιστοιχεί σε κάθε συνασπισμό. Αυτή η υπουργική κρίση δεν αντικατορίζει μόνο την πολιτική κρίση του Λιβάνου. Αφορά επίσης και αντικατοπτρίζει την κοινωνική κατάσταση αλλά και την πνευματική κατάσταση της χώρας. Γιατί δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι λένε οι εφημερίδες. Ε, είναι δύσκολο κανείς να διαβάσει τον τύπο και να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ιδέα για το τι ισχύει στη χώρα γιατί ο τύπος της χώρας ε, όλες, όλες οι εφημερίδες ε, είναι κομματικές, ανήκουν σε κάποιον ασπισμό, στον ένα ή στον άλλο. Οπότε δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσει με την κειμενική ιδέα για την κατάσταση. Κάθε φορά που καθένα διαβάζει ένα άρθρο θα πρέπει να δει ε, η εφημερίδα από την οποία προέρχεται το άρθρο ε, σε ποιον την ιδιοκτησία βρίσκεται. Άρα οι πολιτικές ελίτ ε, δεν, δεν, έχουν κάνει, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, επίσης και οι πνευματικές ελίτ δεν μπορούν να διαχειριστούν την κρίση με επιτυχία. Και δεν σα κρύβω ότι πάρα πολύ δίστασαν να ανταποκριθώ στη σημερινή πρόσκληση. Δεν έχουμε άλλωστε εδώ την ε, Λιβανέζη για την προσωπία ε, για να πει που έχω δίκιο και που έχω άδικο. Όμω, πέραν όλων αυτών, είναι υποχρεωμένοι να κάτσουν και να στήσουν μια κυβέρνηση εθνική ενότητα. κατανομή των πάμε προ εσωτερική αντιπαράθεση και οικονομική κρίση. Είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε πώ θα γίνει η κατανομή των χαρτοφυλακίων, ε, να δούμε ποιο υπουργό θελητη γι' αυτό και τώρα έχουμε το παπαζάρι για τα χαρτοφυλάκια. Υπάρχουν κάποιε ιδιαίτερε, κάποιε ενδιαφέρουσε θέσει που μπλοκάρουν τις διαπραγματευσει ε, πρωτα Πρώτα-πρώτα το χαρτοφυλάκι των τηλεπικοινωνιών και το αντίστοιχο Υπουργείο. Ε, πάρα πολύ επιμαχή θέση. Επίσης το Υπουργείο δικαιοσύνη και επίσης το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας. Παρά όμω αυτή την εμπλοκή, παρά τη δυσπιστία, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει, υπάρχουν κάποιοι όροι και δεν τα ε, παραβιάζει και οπότε συνεχίζεται οι επαφές που παρά το ότι λέγεται ότι είναι μυστικές, στον τύπο πάντα υπάρχουν διαρροές. Σύμφωνα με τη σημερινή δομή, την κυβερνητική, γιατί συνεχίζει και υπάρχει η κυβέρνηση και υπάρχουν ε, υπουργεία που παρά την κρίση συνεχίζουν να λειτουργούν, ε, πάμε προς έναν δεύτερο, ή, ή, θα έχουμε τη σημερινή δομή ή θα έχουμε κάτι άλλο, δηλαδή κυκλική αναλλαγή χαρτοφυλάκια. Ποια είναι τώρα, ποιες είναι οι προοπτικέ ε, διεξόδου από την κρίση. Το να υπάρξει κάποιο είδου επιδιαιτησία. Ε, αυτό θα είναι ένα πρόσωπο που θα συγκεντρώνει κάποιες ε, ιδιότητες. Ε, ας πούμε ότι θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι και επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων που όπως σας είπα αποτελεί σύμβολο εθνικής ενότητας της χώρας. Αυτός θα είναι επομένως ε, διαμεσολαβητής, ούτως ώστε να μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να υπάρξει τελικά κάποια συνεννόηση με βάση κάποιες κοινέ αρχές να αποπολιτικοποιηθεί η προβληματική κατόπιν να τεθούν και να εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες όσον αφορά την κατανομή των, ε, των χαρτοφυλακίων που να γίνει ή αναλογικά με τη δύναμη των πρατάξεων ή με κυκλική εναλλαγή δεύτερη προοπτική των δείξεων από την κρίση. Το να υπάρξει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών που να μην ε, προσανατολίζεται άμεσα ούτε στη μία παράταξη ούτε στην άλλη. Τρίτη λύση διεξόδου. Πολλοί αναλυτές λένε ότι θα πρέπει να αναλύσουμε τη λύση εκτός της χώρας. Γιατί έχουμε αυτή την ε, προσέγγιση με Σαουδική Αραβία και Συρία που θεωρήθηκε από πολλού ε, σαν ένα αισιόδοξο σημείο, ε, σαν αρχή διεξόδου από την κρίση. Για κάποιους Λιβανέζους αναλυτέ, η ΕΠΑ που προγραμματίζονται την κατάσταση σε Ιράκ και Αφγανιστάν έδωσαν την θέση τους εις την Σαουδική Αραβία με την προσέγγιση αυτή που γίνεται και στην ε, Συρία. Στα πλαίσια αυτής της ε, προσέγγισης, κατά τρόπο ηρωνικό, θα βρεθεί, ε, θα βρεθεί κρίση μέσω Δαμασκού. Οπότε έχουμε τώρα αυτούς τους απεσταλμένους που για να έρχονται, ζητείτε κάποια λύση. Ε, ε, γίνεται και συνεννόηση με το Κατάρ, με τη Γαλλία, κάποιο είδου συμφωνία, την Τόχα 2. Και έτσι να βρεθεί διέξω από την κρίση. Εν κατακλείδη θέλω να σας πω ότι παρά αυτό το πεντάμινο της κρίσης συνεχίζει και λειτουργεί η κυβέρνηση και τα Υπουργεία και παρά όλα αυτά ο, ο κόσμος ε, έχει κάποιο είδους ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος και έτσι αγνοεί. Δεν ενδιαφέρεται για τη γενικότερη κρίση. Θα μπορούσε κανείς να βρει μια σύγκριση μεταξύ της βελγικής κυβερνητικής κρίσης και της ε, λιβανέζικης. Πάντοτε τα δελτία ειδήσεων ξεκινάνε με, με τον κακό καιρό, κάποιο είδου ε, καταιγίδε, πλημμύρε κλπ. Και μετά ε, αρχίζει η αναφορά στο κάθε στρατόπεδο, στην κάθε συμμαχία. Σα ευχαριστούμε κύριε Σφαίρα, ευχαριστούμε και για την υπομονή σα, λέει πρόεδρο. Όπω προαναφέραμε, δεν θα υπάρξει ανταλλαγή σε μια που ε, δεν είναι εδώ η Λιβανή για την προσωπία. Οπότε, θα υπάρξει η ευκαιρία να επανέλθουμε στα του Λιβάνου σε άλλη συνάντηση με την παρουσία των ε, Λιβανέζων συναδέλφων. Και τώρα συνεχίζουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι ε, μπορείτε να αποχωρήσετε. Euh, euh, να σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 6. Ανταλλαγή απόψεων για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κάλσον, τον συντονιστή Euromed, ο οποίος εκπροσωπεί την Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ένωση για τη Μεσόγειο γιόρτασε την πρώτη της επέτειο στις 13 Ιουλίου του 2009. Όπως θα το γνωρίζετε, λόγω της στρατιωτικής παρέμβασης του Ισραήλ στη Γάζα, οι συνεδριάσεις του εκτελεστικού τμήματος της Ένωσης για τη Μεσόγειο μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου αναβλήθηκαν. Οι εργασίες στη συνέχεια συνεχίστηκαν σε επίπεδο υψηλών ύπατων ε, υπαλλήλων και υπουργών. Επίσης οργανώθηκε αποστολή ε, στο Ισραήλ, την Γάζα και την ε, περιοχή του τη Λωρίδα της Γάζας στον εκτάκτος και επίσης οργανώθηκε και η πρώτη υπουργική συνεδρίαση για την Ένωση της Μεσογείου για την βιώσιμη ανάπτυξη ασχολήθηκε η σε αυτή με τέσσερι βασικές προκλήσεις για το περιβάλλον. Το νερό, τις μεταφορές, την ενέργεια και την αστική ανάπτυξη. Έπειτα στις 7 Ιουλίου στι Βρυξέλλες οργανώθηκε συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ένωσης για το Μεσόγειο στα περιθώρια του ΕΚΟΦΗΝ. Η συνεδρίαση αυτή ήταν ευκαιρία για να συζητηθούν η οικονομική κρίση και να γίνει συζήτηση με την παρουσία της Σουηδικής Προεδρίας. Έπειτα συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών τη Ένωση για τη Μεσόγειο που προβλεπόταν για τι 24 και 25 Νοεμβρίου στην, ε, στην Κωνσταντινούπολη. Ακολουθεί άλλε δύο υπουργικέ συνεδριάσει ε, για τον Νοέμβριο. Ενίσχυση του ρόλου των γυναικών ε, στην κοινωνία, στο Ραμπάτ στι 11 και 12 Νοεμβρίου και συνεδρίαση για το περιβάλλον στο Ντουμπρόβνικ στι 25 και 26 Νοεμβρίου. Έπειτα, υπουργική συνεδρίαση για το εμπόριο στις 9 και 10 του μήνα στις Βρυξέλλες. Όπως σας έλεγα συνάδελφοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον συντονιστή για την Euromed, τον κύριο Κάλσον και από διοικητική πλευρά ελπίζω ότι θα μας ενημερώσετε κύριε Κάλσον για τη συνέχεια των συζητήσεων που αφορούν τη δημιουργία τη γραμματείας, του οποίας το καθεστώ θα πρέπει να εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση, είπα των υπαλλήλων στις 23 Νοεμβρίου και από πολιτική σκοπιά ελπίζουμε ότι θα μας δώσετε κάποια στοιχεία για το πώς θα εξακολουθήσει η συνεργασία των Υπουργών Εξωτερικών και η συνεδρίασή τους που προβλεπόταν στις 24 και 25 Νοεμβρίου και η οποία δεν θα γίνει. Ε, ίσως έχετε λοιπόν πληροφορίες να μας πείτε. Κύριε Κάλσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Με χαρά έρχομαι να σας ε, μιλήσω για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μεσογείου. Εφόσον έχουμε και την τιμή ως χώρα να προεδρεύουμε μέρο μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα πολύ σαφές όραμα ως προς την ευρωμεσογειακή διάσκεψη. Είναι η γειτονία μας αυτή και έχουμε και σαφές όραμα για τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τις υποχρεώσεις μας ως προεδρεύοντων ή ε, συμπροεδρευόντων στην διαδικασία αυτή. Ξέρετε ότι έχει αναπτυχθεί η Ευρωμεσογειακή Ένωση μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όμως ε, εμείς δεν διστάσαμε ποτέ ως προς τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει μέσα από τις ε, κοινέ διακηρύξεις Παρισίων και Μασαλίας. Και πριν προχωρήσω, Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω, να αποτείνω μάλλον ε, φόρο τιμής ε, στις, ε, στις προεδρίες της ΕΜΠΑ και στην περίοδο της κρίσης στη Λόρδια της Γάζας και στη στάση γενικά που έχει τηρήσει την υπόθεση αυτή, ιδιαίτερο στην επίσκεψη 25 Φεβρουαρίου εφέτος. Επιπλέον, είχαμε την συζήτηση της κατάστασης, την αντιμετώπιση της κατεπίουσας ε, ανάγκης σε μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη. Κυρία Πρόεδρε. Ύστερα από την επανάληψη των δραστηριοτήτων μόλις επτά ημέρες αφού το αναλάβαμε την ε, Προεδρία εμείς, Περάληψη λοιπόν διαπραγματεύσεων ε, και επαφών με υπουργού οικονομία και οικονομικών προσπαθούμε να αναλάβουμε τις, ε, να προωθήσουμε μάλλον τις επαφές, την υλοποίηση των επαφών και διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο και κυρίως στο πολιτικό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε πρόοδο ως προς το καθεστώς της ε, γραμματείας που θα εγκατασταθεί στην θα εδρεύει στη Βαρκελόνη, έτσι ώστε να ξεκινήσει το χειρότερο δυνατό η εργασία αυτού του σώματος με βάση την πρόοδο που έχουμε ήδη επιτύχει. Τομείς πολύ σημαντικοί για την περιοχή, ασφαλώς, θα έχουν να κάνουν με την ρήπανση των θαλασσών, τις υποδομές, τις μεταφορές, τις εναλλακτικές πηγές ε, ε, ενέργειας, ε, την ανώτερη εκπαίδευση, τομείς που θα δράσουν καταλητικά και για τις επενδύσεις που θα προσελκύσει η περιοχή και που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε περισσότερη εμπιστοσύνη, ανάπτυξη εμπιστοσύνη στην ε, περιοχή. Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά πρόεδρε, ελπίζουμε και σκοπεύουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία στις 23 Νοεμβρίου. Θεωρούμε ότι είναι ασφαλές, ασφαλής πρόγνωση το να περιμένουμε ότι θα έχουμε καλή πρόοδο και εξέλιξη με την συμβολή όλων των πλευρών, με την ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ε, γείτονες της Μεσογείου. Τόσο εμείς όσο και οι μεσογειακοί εταίροι έχουν ως βασικό πρόβλημα, έχουμε ως βασικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε τη ρήπανση και πρέπει να πω ότι δεν είναι ισότιμη η κατανομή του προβλήματος. Πρέπει επίσης να καταβάλουμε κάθε την προσπάθεια για να προαγάγουμε την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Να εξασφαλίσουμε το ότι οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν ε, θα οδηγήσουν σε χάος και αποσταθεροποίηση. Τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε όλοι, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Και χρειαζόμαστε όλοι περισσότερο διάλογο και συνεργασία. Επίσης, υπάρχουν ε, και άλλοι τομείς στους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα στην ε, περιοχή μας. Σε παράδειγμα, τη συζήτηση του ρόλου των γυναικών στις κοινωνίες μας, άλλο ένα πρόβλημα κρίσιμο, στο οποίο χρειάζεται συνεργασία μας. Και ένας άλλος ε, τομέας, πολύ σημαντικός επίσης, είναι οι διαπολιτισμικές σχέσεις. Η διαδικασία της Βαρκελόνης έχει ήδη εντοπίσει, αναγνωρίσει σημασία αυτής της συνεργασίας μέσα από το ενίδρυση του Ιδρύματος Αναλίντ, στο οποίο συμμετέχουμε όλοι κατά τρόπο επικοδομητικό, πιστεύω. Η αμοιβαία κατανόηση, η αμοιβαία ε, συνεννόηση είναι καλύτερο τρόπος να αντιμετωπίσουμε του εξτρεμισμού κάθε είδου. Η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι έχουν ασφαλώς πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν προκειμένου. Πρόεδρε, η συνάντηση των Υπουργών στην Κωνσταντινούπολη, όπω είπατε, χρειάστηκε να αναβληθεί, αλλά γνωρίζουμε ασφαλώ ότι ε, δεν είναι η στιγμή τώρα, μάλλον το κλίμα τώρα, πρόσφορο για τέτοιου είδου συνάντηση. Εργαζόμαστε σκληρά για να προετοιμάσουμε τρει ε, τομεακού χαρακτήρα υπουργικέ ε, συναντήσει που αναφέρατε και εσεί, Πρόεδρε, για τι επόμενε εβδομάδε. Είχαμε την πρώτη συνάντηση τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες, μετά έχουμε άλλη μία που προβλέπεται για τους υπουργούς υπεύθυνου για θέματα γυναικών, το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, που προβλέπεται να διεξαχθεί στο Μαρακέ στι 11 και 12 Νοεμβρίου. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ε, συνεδριάζουν στο Κάιρο οι δικοί μας ε, για να επεξεργαστούν το κείμενο που θα υποβληθεί προ έγκριση στην συνεδρίαση αυτή. Επίση, προπαρασκευή βρίσκεται και μια ε, συνεδρίαση για τις 26 και 27 Νοεμβρίου στο Μπρόβνικ σε θέματα περιβάλλοντος ε, με μελέτη του της, προόδρου, της προόδου με θέματα του ορίζοντα 2020 20, και διάφορες ε, και προτάσεις για την ε, για κοινή διακήρυξη θέσεων Ένωσης για τη Μεσόγειο. Επίσης θα γίνει αργότερα στις Βρυξέλλες σε 9 Δεκεμβρίου συνεδρία των Υπουργών Εμπορίου με ορίζοντα το 2010 που μας περιμένει και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Έχουμε κύριες προτεραιότητες λοιπόν, αυτές εδώ τις συνεδριάσεις σας ανέφερα ως Προεδρία και μαζί με την σύσταση της ε, Γραμματείας και την ε, υιοθέτηση του καθεστώτος της Γραμματείας μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει τους στόχους μας, τους κύριους στόχους της Προεδρίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα για τη γραμματεία να υποβάλω απευθεία μια ερώτηση. Είπατε ότι θα εγκριθεί το καταστατικό της. Ε, για το γενικό γραμματέα Για γενικό γραμματέα έχετε κάποιο πρόσωπο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για την εκλογή γενικού γραμματέα στην ε, συνεδρίαση των υποτανοικοσόπων τον Σεπτέμβριο, στις 30 Σεπτεμβρίου αν σωστά θυμάμαι, οι συμμετέχοντες, οι εταίροι μας, προσκλήθηκαν να υποβάλουν υποψηφιότητες για αυτές τις θέσεις. Και επειδή η έδρα της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα βρίσκεται στη Βαρκελόνη, στην βόρεια ακτή της Μεσογείου. Υποθέτουμε ότι η Γενική Γραμματεία μάλλον θα προέρχεται από την νότια πλευρά της Μεσογείου. Στην ε, συνεδρία του Σεπτεμβρίου κάναμε λοιπόν αυτήν την έκκληση να υποβληθούν υποψηφιότητες προς την Προεδρία. Ως τώρα όμως έχουμε έχουμε μόνο έναν υποψήφιο. Μία υποβολή υποψηφιότητα. Ο στόχο μα, είναι να διορίσουμε Γενικό Γραμματέα στη συνάντηση της 23 η Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε κύριε Κάρλσον. Οπότε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέντουμι. Είχατε παρέμβει και το πρωί. Τον είχατε ζητήσει. Όχι. Όχι τώρα. Ωραία. Πάντως το λόγο σας τον έδωσα. Ο κύριος Σαντούκα. Σαντούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, πρόσωπο της Προεδρίας για όλες τις ιδέες που συνεισέφερε στο θέμα της Ένωσης της Μεσογείου. Και χαίρομαι που βλέπω ότι τα εμπόδια, οι φραγμοί για τη διαδικασία προέρχονται από τα θέματα της Γάζας βέβαια και της ευρωτικής παρέμβασης εκεί και των εξελίξεων στην περιοχή. Όπως θα θυμάστε η διαδικασία της Βαρκελόνης είχε και άλλα εμπόδια, είχε παρόμοια εμπόδια, αλλά χρειάστηκε να τα ξεπεράσει. Παρ' όλα αυτά δεν οδηγήθηκε σε αίσιο πέρας ε, με όλες αυτές τις συγκρούσεις. Ένα από τα σχόλια που έκαναν πολύ επίσημη σε ανώτατο επίπεδο και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση με τα σχόλια του Πρόεδρου Σαρκοζή επεσήμαναν ότι οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν κυρίως στις οικονομικές πτυχές και όχι τόσο στις πολιτικές και στην πολιτική συνεργασία. Θα μπορούσα λοιπόν και εγώ να πω ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί αν παραμελούμε τους πολιτικούς παράγοντες ο πολιτικό παράγων είναι ο σημαντικότερο για την επιτυχία μια οποιασδήποτε τέτοια διαδικασία, μια διεθνού πρωτοβουλία. Ελπίζω λοιπόν ότι τα διδάγματα της διαδικασίας της Βαρκελόνης θα μας επιτρέψουν να βρούμε την κατάλληλη λύση στη σημερινή κατάσταση. Ελπίζω λοιπόν για όσους θέλουν να επιδιώξουμε μόνο οικονομικούς στόχους χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το πολιτικό σκέλος να μην παραβλέπουν τι συνέβη στην περιοχή μας την τελευταία χρονιά. Επηρεάστηκαν τα βήματα που είχαν σχεδιαστεί και διαδικασίες που έπρεπε να έχουν ξεκινήσει ήδη δεν έχουν προχωρήσει. Ελπίζω λοιπόν ότι για τις μελλοντικές μας προσπάθειες θα, έχουμε, θα βασιστούμε σε αυτή την πρόσφατη εμπειρία. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για την κατάσταση της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορεί το ζήτημα αυτό να το παραβλέπουμε. Πρέπει να έχουμε πίστη στο ότι μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο στα οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ενώ οι διμερείς ε, μορφές συνεργασίας μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου, της Βόρειας και της Νότιας, θα, προχωρά, θα προχωρεί. Ε, δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι δεν πρέπει να παραβλέπετε το ζήτημα τη Παλαιστίνης, εάν θέλουμε θετική μορφή συνεργασία μεταξύ των χωρών τη λεκάνη τη Μεσογείου. Όποιο τίτλο και δώσουμε σε αυτήν την ε, διαδικασία συνεργασία Ένωση για τη Μεσόγειο, διαδικασία τη Βαρκελόνη ή οτιδήποτε. Αυτό είναι μια πρόσκληση προς τους συναδέλφους από την βόρεια ακτή της Μεσογείου και από όλες τις μεσογειακές χώρες να επιδιώξουν αυτόν τον κοινό στόχο. Είτε θέλουμε, μάλλον εάν θέλουμε πραγματική και αυθεντική σταθερότητα και ειρήνη και συνεργασία για όλους τους τομείς, σε όλες τις χώρες, αυτό δεν θα το πετύχουμε ποτέ εκτός και δώσουμε τέλος στην σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών, Αράβων και Παλαιστινίων. Και αν δεν θέσουμε τέρμα στην Ισραηλινή κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών. Σας θυμίζω ότι αυτή είναι η τελευταία υπάρχουσα κατοχή, η τελευταία πραγματική κατοχή στη σύγχρονη εποχή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σαντούκα. Παρακαλώ. Από την Τινησία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Και δεν μπορώ παρά να πω το καλώς σε όλους εδώ που ήρθαν από τη χώρα μας ε, αμέσως μετά τις πρόσφατες εκλογές, όπως ξέρετε εμείς, ανέκαθεν ε, έχουμε ε, ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα για την ευρωμεσογειακή υπόθεση και πάντοτε θεωρούμε ότι όλα αυτά ωφελούν για την ευημερία και την ειρήνευση στην ε, περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, η σημερινή μας συζήτηση πρέπει να τύχει κάποιε ιδιαίτερε προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε αυτό το οποίο συζητούσαμε σήμερα το πρωί. Συζητούσαμε το θέμα τη ειρήνη, τη ειρήνευση στην Μέση Ανατολή, αλλά και τη ευημερία εκεί και όπω προείπε ο συνάδελφο. Ε, έχουμε θέμα ε, επιρροής της ε, διαδικασίας της Βαρκελόνης και η Τινησία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του θεάτρου, αυτής της σκηνής ε, της Ευρωμεσογειακής. Και ανέκαθεν ήμασταν ε, καλοί γείτονε στην Ευρώπη, ήμασταν ότι ε, αναφαντών υπέρ οποιασδήποτε πρωτοβουλία για συνεργασία και ευημερία στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, δεν κατάλαβε ο λαός μας κάποιο είδους θετική επίδραση, κάποιο είδου πρόοδο και ιδίω μιλώ για τους νέους. Εμείς εκπροσωπούμε το λαό μας. Εμείς παρακολουθήσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κάλσον, τον οποίο και ευχαριστούμε γιατί επιδεικνύει τόσο ενδιαφέρον για τα θέματά μας ε, κάποιος ο οποίος ε, προέρχεται από την Σκανδιναβία. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι φραγμοί ποια είναι τα εμπόδια στην ε, πρόθεση της υπόθεσης της, ε, της Βαρκελόνης. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ώστε απρόσκοπτα να συνεχιστεί αυτή η πορεία που ξεκίνησε και όπως προαναφέρθηκε να μην λησμονούμε ότι αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Μεσόγειο. Όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα πρετανεύσουν τα πολιτικά κριτήρια και όχι τα οικονομικά. Να δούμε δηλαδή πρώτα πώς έχει πολιτική συγκυρία και κατόπιν η οικονομική. Πάντως ε, όλα αυτά τα μέτρα, στις πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ θετικά και φυσικά και είναι αντίστοιχες των προσδοκιών που υπάρχουν. Να λάβουμε υπόψη ότι στο Νότο σήμερα η νεολαία έχει κάποιες προσδοκίες. Θέλει να ζει υπό τις ίδιες συνθήκες όπως και η νεολαία στον Βορρά. Γι' αυτό και εμείς και ο πρώτος Μπενάλη συγκεκριμένα αντίστοιχη πολιτική ασκούμε για την νεολαία και γι' αυτό και προσχωρήσαμε στην ιδέα ε, του έτους της νεότητας οπότε νομίζουμε ότι η Ευρωμεσιακή Διάσκεψη θα πρέπει να βάλει το λιθαράκι της στην υπόθεση αυτή. Το 2010 επομένω να είναι ένα πετυχημένο έτος για την νεολαία και πιο συγκεκριμένα για τη νεολαία της Μεσογείου. Και εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλες οι προσδοκίες του λόγου μας για, αυτό το, για αυτή την ιδέα. Οπότε κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται θα πρέπει να είναι αντίστοιχη. Νομίζω ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα δεν αντιστοιχεί στις προσδοκίες και νομίζω ότι και οι συναντήσεις μας ίσως δεν είναι αντίστοιχες τη ε, της σημασίας που έχει αποδοθεί ε, από όλους μας ε, στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης ε, για την νεολαία. Καθέσει πλέον. Λοιπόν. Εμείς προσπαθήσαμε να ανανεώσουμε την εικόνα της χώρας. Και όσον αφορά επίσης την αντίληψη για την συνεργασία Βορρά και Νότου. Να δούμε, προσπαθήσαμε, πώς θα έχουμε αναβάθμιση της ε, θεσμικής επικοινωνίας. Να υπάρχει περισσότερη ελευθερία, να αναπτύξουμε περισσότερο την, τον κοινωνικό μας βίο. Ε, τροποποιήσαμε ένα νομοθετήματα της χώρας. Ε, φροντίζουμε να δούμε πώς θα τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. πώς με κάθε τρόπο θα βοηθούμε στην βελτίωση των σχέσεων βορανότου. Θέλουμε να έχει γίνει αποτελέσμα τη και διάσκεψη και θέλουμε, όπως προαναφέρθηκε σήμερα το πρωί, να είναι η Επιτροπή μας ένα βήμα νυφάλιο και αξιοπρεπούς διαλόγου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συντονιστή, τον κύριο Κάλσον, για την σύντομη αυτή παρουσίασή του, για τις διάφορες δραστηριότητε που ετοιμάζονται από ευρωπαϊκέ. πλευρά. Να του θέσω κάποιε ερωτήσεις, αν μου το επιτρέπει. Κατά πρώτον, δεν γνωρίζω εάν η σύγκρουση Ισραηλινών και Αράβων που δεν έθιξε. Είναι μια από τις προτεραιότητε της Προεδρίας. Νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία για τον ευρωμεσογειακό χώρο αυτό. Έπειτα, ένα ακόμα ερώτημα. Η κοινοβουλευτική συνέλευση της Euromed. Εδώ δεν θέλω να αναπτύξω το σημείο αυτό, γιατί θα το δούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διαταξή με λεπτομέρειε, αλλά εκείνη τι ε, έχουν προβλέψει. Έχουν προβλέψει κάτι ώστε η συνέλευση αυτή να γίνει όπως συχνά ζητήθηκε η κοινοβουλευτική διάσταση της Ένωσης για την ε, Μεσόγειο. Και τέλος, κύριε Κάλσον, μιλήσατε για το καθεστώς της δραματείας. Υπάρχουν δυσκολίες ή προβλήματα κατά τις διαπραγματεύσεις. Τι μέλη γενέστε με αυτό το καθεστώς Ευχαριστούμε κύριε Μεσκή. Ο κύριο Αντάντ από τη Συρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ίσως να μην έχω τίποτε το σημαντικό να προσθέσω στα όσα είπε ο Παλαιστίνος την ο Αλγερινός συνάδελφος. Αλλά πολύ σύντομα επιτρέψτε μου να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε μπορέσει να ε, ολοκληρώσουμε την διαδικασία τη σχετική με το καθεστώς. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ξεκίνησαν την εποχή της επιθέσεως των Ισραηλινών κατά της Λωρίδας της Γάζας. Και εκεί αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την ε, Στι συναντήσει ει ένδειξη διαμαρτυρία. Αυτό που ζητούμε από του Ισραηλινούς είναι ο σεβασμό τη δικασία Βαρκελόνη, των εταίρων του, του ανθρωπιστικού δικαίου. Συναντήσει και συστήσει μπορούν να γίνονται. Όπως και έγιναν και συνεχίστηκαν το 2009 με την γαλλο-αιγυπτιακή ε, διακήρυξη για τη συνέχιση των προσπαθειών, την οποία ακολούθησαν και άλλες ε, δηλώσεις ε, με αποτέλεσμα ε, αραβικά κράτη να αποχωρήσουν από τις ε, συναντήσεις, από τις συνεδριάσεις. Οι προσπάθειες, όπως υπόθηκε από τους προελήφθαντες, ήταν πολύ περιορισμένες. από, όλες τις, από τους κύριους ε, παράγοντες, λίγες είναι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν στην ε, διαδικασία επίλυσης της Αραβο-Ισραηλινής διαφοράς. Ακόμα παραμένουν δε ως προς την ε, γραμματεία εκκρεμότητες όπως ο ορισμός του προσώπου του Γενικού Γραμματέα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιος είναι, πρέπει να συζητηθεί το θέμα να είναι ο Γενικός Γραμματέας ικανός να κρατήσει τη θέση αυτή. Εμείς άλλωστε έχουμε καταγράψει μια προκατακτική συμφωνία σχετική με θέματα χρηματοδότησης, ενέργειας κλπ. Αλλά ακόμα δεν έχουν ρυθμιστεί θέματα που αφορούν άλλες θέσεις. Έχουν ε, εκφραστεί όμως αντιδράσεις εντωμεταξύ ε, από τα αραβικά κράτη, παραδείγματι στην υποψηφιότητα Εβραίου ε, για τη θέση του Αντιπροέδρου, για τα θέματα της εκπαίδευσης από τον Λίβανο. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει η θέση που θα αντιστοιχεί στο Ισραήλ να ε, μην ε, δοθεί, να μην υπάγεται σε τομείς κρίσιμους για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ήταν πολλοί οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν σε επιβράδυνση διαπραγματεύσει και σε αποτυχία την προσπάθεια εξέβρεση συμφωνίας. Η ευρωπαϊκή πλευρά, άλλωστε, βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίζει με αρκετή σοβαρότητα την ε, κατάσταση, την πολιτική κρίση που έχουμε, όπως άλλωστε επιθυμούν και οι Ισραηλινοί. Από την άλλη πλευρά, πολλά είναι τα αραβικά κράτη τα οποία επιμένουν πρώτα απ' όλα να διεξαχθεί ο πολιτικός διάλογος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πελιό, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια απορία ως προς τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε το ρόλο της ε, ε, Ένωσης για την ε, Μεσόγειο. Εάν θεωρούμε ότι το τεράστιο αυτό εγχείρημα Ένωση για τη Μεσόγειο εγχείρημα και σχέδιο το οποίο μας πηγαίνει πολύ μακριά στο μέλλον ελπίζω ε, πρέπει για να αρχίσει να εργαζεται, να λειτουργεί να έχει προηγουμένως επιλύσει την αραβο-ισραηλινή ε, σύγκρουση προφανώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το δούμε να υλοποιείται έχουμε όπως γνωρίζετε ασφαλώς μεγάλη εμπειρία από αδελφοκτόνους πολέμους. Το πρωί ακούστηκε και ο όρος ολοκαύτωμα. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικά ξεκινά, έχει σαν στάση να ξεκινά από συγκεκριμένε πρωτοβουλίε, όπω για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, και προτάσει συγκεκριμένε με συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία από ό,τι άκουσα και το πρωί κάποιοι αποκάλεσαν συγκεκριμένε πρόοδου, το είπε ο κ. Σαμπτουλά, ε, με συγκεκριμένη δηλαδή πρόοδο που καταμετρήσιμη, μετρήσιμη πρόοδο. Και ίσως αυτό που δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε διπλωματικά με τις πολυμερές διαπραγματεύσεις εδώ και 18 χρόνια θα ήταν καλό να μην αποτελέσει και το λόγο αποτυχίας της Ένωσης για την Μεσόγειο. και να καταδίσουμε τελικά τα κράτη της Ένωσης που θα μπορούσαν να είναι μέλη της Ένωσης να περιοριστούν σε διμερείς σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ με διακυβεύματα τεράστια σημασία για την Ευρώπη, μεν, αλλά κυρίω για την νότια όχθη τη Μεσογείου και για τι σχέσει με την Ευρώπη. Και πάνω απ' όλα απαραίτητο είναι η πολυμερής προσέγγιση και γι' αυτό θεωρώ ότι η πολιτική μας κοινοβουλευτική ε, επιτροπή θα πρέπει ξεκάθαρα να ε, δηλώσει τη βούλησή της για συνέχιση σε αυτό το πολιτικό οικοδόμημα, ακόμη και όταν πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να συνεχίσει. Ξέρουμε ότι ο καθένας έχει τις δικές του προτεραιότητες και προτιμήσεις, αλλά όταν είμαστε εμείς εδώ από τις διόχθες της Μεσογείου βουλευτές, πρέπει κύριο μας μέλημα να είναι η Ευρώπη που πολλά έχει να κάνει και πολλά μπορούμε, μπορεί να προσφέρει να βοηθήσει και να προχωρήσουν οι σχέσεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Όχθης έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε μια ατέρμονη ουσιαστικά ομοιρία δηλαδή την Άραβο-Ισραηλινή σύραξη. Βεβαίως θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε υπέρμαχοι του ή όλα ή τίποτα ε, και ακούω με προσοχή και τα λόγια όσων λένε ότι θα πρέπει να λησμονηθεί το θέμα αυτό δεν πρέπει να μπει στο περιθώριο, όπως άλλωστε έγινε τον Ιούλιο. Ε, το να λέμε όμως ότι είναι προτεραιότητα φυσικά είναι αυτονόητο, δεν μπορεί όμως και να σημαίνει ότι η Ένωση για την Μεσόγειο μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν λυθεί η αραβιστρολινή διαφορά. Για την νεολαία Υπάρχουν προβλήματα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν προβλήματα. Στη βιώσιμη ανάπτυξη υπάρχουν προβλήματα. Ε, λοιπόν, α προχωρήσουμε με αργά και σταθερά βήματα. Μια μέθοδο την οποία ε, χρησιμοποίησε με αποτελέσματα πολύ θετικά η Ευρώπη, όχι πριν από τρει αιώνε, αλλά μόλι πριν από 50 χρόνια και μπόρεσε να έχει σαφή πρόοδο και αποτελέσματα. Α κάνουμε λοιπόν ευφυεί επιλογέ και α μην μετατρέψουμε ε, σε σημείο κλειδί την αραβο διένεξη με αποτέλεσμα τελικά να αποτύχουμε σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σταμπάρκη, έχει το λόγο από την Τινησία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι όντω πολύ σημαντικό το θέμα. Και πιστεύω ότι αυτά που είπαν οι συνάδελφοι από την ε, νότια όχθη της Μεσογείου έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε λίγο πολύ με το βάπτισμα του πυρός για την ε, Ένωση για τη Μεσόγειο. Ο βάρος του πυρός ήταν δηλαδή η επίθεση εις βάρος της Λόρας της Γάζας. Ένα τραγικό διαστάσεων γεγονός που ασφαλώς δεν μπορεί κανείς να λησμονήσει από τη μια μέρα στην άλλη. Και έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες εμείς ιδιαίτερως από την Τινησία, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ανήγγειλε τέτοιο σημαντικό ε, εγχείρημα ο πρόεδρος Σαρκοζή. Όλοι έχουμε υποστηρίξει αυτή ε, το, αυτό το εγχείρημα, αυτή την πρωτοβουλία. Όμως οι εξελίξεις δείχνουν ότι ο πολιτικός τομέας, ο, η πολιτική επηρεάζει τις δομές και ή την ανάπτυξη νέων δομών και ό,τι και να πούμε ως προς τον πολιτικό τομέα, οι άλλες διαστάσεις του ε, οι άλλε διαστάσει του πολιτικού προβλήματο ε, των προβλημάτων δεν μπορούν να επιληθούν εφόσον δεν επιληθούν τα πολιτικά προβλήματα. Πάντα θα επηρεάζονται δηλαδή όλοι οι τομεί από τα πολιτικά, την πολιτική πτυχή. Είπατε κι εσείς ότι από την θέσπιση της Ένωσης έχουμε επιτύχει μέσα σε ένα χρόνο την ε, δραστηριοποίησή μας για περίπου ένα εξάμεινο και την αδράνεια για ένα περίπου τετράμινο μετά, λόγω των γεγονότων τις οποίες έγινε ο δινηρός μάρτυρας η Γάζα. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Κάλσον σε ποιο βαθμό έχουμε προχωρήσει εδώ έχουμε μιλήσει για ζωτική σημασία σχέδια για την περιοχή, για την ανάγκη για ανάπτυξη της, ε, των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των δύο όχθεων, για την ανάγκη να προστατευτούμε από τη ρήπανση. Τι έχουμε επιτύχει από όλα αυτά λοιπόν. Τι έχουμε επιτύχει και ως προς την πολιτική προστασία και ως προς την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ως προς την ε, ενεργειακή τεχνολογία. Επίσης ε, για την οικονομία θα ήθελα να αναφερθώ στην μεγάλη οικονομική κρίση η οποία έχει συγκλονίσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τις λάβω τόσο πολύ υπόψη μου εδώ γιατί απέχουν πολύ από την Ευρώπη και την Αφρικανική Ήπειρο. Έχει επηρεάσει λοιπόν ε, δεινά η χρηματοπιστωτική κρίση στην οικονομική μας κατάσταση, γιατί είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα στις χώρες μας. Και... Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει, όπως είχε συζητηθεί πριν από δύο χρόνια στην Τινησία, να συζητηθεί το θέμα της ε, ανάπτυξη της Κεντρικής Τράπεζας για την ε, Ευρωμεσογειακή Συνεργασία. Αυτό το εγχείρημα έχει λησμονηθεί μάλλον. Δεν έχουμε ακούσει τίποτε για πρόσφατες εξελίξεις ή αποφάσεις από την Τινησία και μετά. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε κύριο Σομπιόλς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όσα μας εξήγησε ο κ. Κάλσον από πλευράς ειδικέ Προεδρίας ήταν πάρα πολύ χρήσιμα διότι η περιγραφή του ε, ήταν περιγραφή που περιορίστηκε στα πραγματικά περιστατικά αυτής όλης της πορείας, της ολοκλήρωσης της ευρωμεσοϊκής συνεργασίας και τα τελευταία χρόνια. Οπότε και εμείς τώρα με τρόπο αμερόληπτο έχουμε μια φωτογραφία, μια απεικόνηση μπροστά μας του πώς έχει η σημερινή κατάσταση. Και κατά τη γνώμη μου η κατάσταση αυτή ε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράδοξο όσον αφορά την αρχική σύλληψη αυτού του οράματος και όσον αφορά ε, αυτή την πρώτη εμπειρία από την πρώτη διαδρομή. Γιατί αν κατάλαβα καλά από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βασική πρόταση ε, της Ευρωμεσογειακής Ένωσης σε σχέση με αυτό το υπήρχε προηγουμένως, δηλαδή η διαδικασία του, του, της Βαρκελόνης που ξεκίνησε το 1995 ε, πρόκειτο για κάτι λέγω το οποίο είχε ως θεμέλιο δύο ιδέες ε, πρώτα-πρώτα μια αποπολιτικοποίηση της ε, ευρωμεσογειακής σχέσης και επομένως πρόκειται για μια πιο λειτουργική σχέση ε, ακριβώς όπως τα εξήγησε ο συνάδελφος Βενσάν Παιδιών όσον αφορά κάποια μεγάλα σχέδια και προγράμματα. Την άλλη μεριά, μια θεσμοποίηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων μέσω ε, της ε, συγκρότησης, της μόνιμης γραμματείας και μιας δομής πιο κεντροκατευθυνόμενης. Οπότε από την πρώτη φάση στη δεύτερη ε, έγινε η μετάβαση που χαρακτηρίζεται όμως από, αυτό το παράδοξο που είπα διότι στην πρώτη φάση η διαξίδη Βαργελόνης ήταν κάτι σαν δίκτυο διμερείς σχέσεις μεταξύ ε και κάποιες άλλες χώρες μιας ιονή μιας τρίτης χώρας. Γιατί λειτουργούσε με δίκτυο και παρά κάποια τραγικά συμβάντα συνεχιζόταν αυτή η σχέση με αυτή τη δομή. Τώρα έχουμε μια πιο θεσμοποιημένη ε, σχέση, δομή, πιο ε, έφτακτα ιεραρχημένη. Οπότε αυτή η τραγωδία της Γάζας δεν επέφερε παράλυση. Και είδαμε καλά από την άλλη μεριά ότι επέφερε ε, μία τροχοπέδη, μία επιβράδυνση της ε, ολοκλήρωσης. Επομένως, εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε το πώς θα προχωρήσουμε προς μία άρση του παράδοξου και της αντίφασης. Μπορούμε επομένω να κάνουμε τα εξή. Πρώτον, να προχωρήσουμε προ μια αποπολιτικοποίηση των σχέσεων αυτών και να στηριχτούμε σε οικονομικέ σχέσει, λογιστι... ε, λειτουργικέ σχέσει, ε, ε, σχέσει επιμελητία του ΣΥΠΗΝ. Άρα, ολοκληρωτική αποπολιτικοποίηση δεν είναι ποτέ δυνατή, αλλά όσο γίνεται περισσότερο. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε δεσμευτεί του να αποκτήσει και πολιτικό υπόβαθρο η Ένωση για την Μεσόγειο. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ εδώ 100% με τα όσα είπε ο συνάδελφος Τελπίκια. Που είπε ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε τις διακηρύξεις για τα μεγάλα λόγια και να έχουμε κάποιες στέρεες τοποθετήσεις ε, που να χαρίζονται από ομοφωνία, από ευρεία μειοψηφία για το διάλογο, για την ειρήνη και για την άρση αυτών των φραγμών που έχουν μέχρι τώρα εμποδίσει το να τον αναδειχθεί αυτός ο ορίζον που επιθυμούμε της ευημερίες και τις ειρήνες και από την άλλη μεριά, όπως είπε και ο Πεγιόν, να κάτσουμε και να δούμε ότι όσο και να θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποια ειρηνευτική συμφωνία, να μην ξεχνούμε ότι αυτός ο στόχος είναι κάτι το δύσκολο, κάτι το ε, πολύπλοκο και επομένω η πορεία αυτή θα είναι αργή, βραδία. Με αυτό να το ξέρουμε, ενώ ταυτόχρονα προχωρούμε. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να τα κουκουλώνουμε αυτά τα προβλήματα και να προχωρούμε την άλλη μεριά σε κάποια προγράμματα και, και, και έργα, δηλαδή κουκουλώνοντας την ε, Παλαιστινο-Ισραηλινή κρίση. Συντοποιώντας το από την άλλη μεριά, είναι θετικό αυτό το στοιχείο και ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να βάζουμε λιθαράκι μας, ώστε να έχουμε μια μια, μια, μια διευκόλυνση της ε, επίλυσης του Παλαιστινιακού. Εδώ δεν έχουμε αντινομία, έχουμε στόχους που συγκεράζονται. Απολυτικοποίηση επομένως. Λειτουργική απολυτικοποίηση, που δεν είναι 100% δυνατή. Απλώς να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο μια πολιτικοποίηση που να φτάνει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να, να μην παραλύει όλο το σύστημα με το παραμικρό πρόβλημα. Και έτσι να ανατενίζουμε, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τη ε, Μεσογείου, τόσο ώστε να μην φρενάρουμε και να συνεχίζεται αυτή μα η πορεία προ την υλοποίηση των οραμάτων μα. Κύριε Μπιόλ, σα ευχαριστούμε και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπεντουμή, εάν είναι έτοιμο να λάβει το λόγο για την Αλγερινή αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την αραβική γλώσσα για να χαιρετήσω, σαλαμαλέκουμ, και μετά να περάσω στα αραβικά και στην υπόλοιπη παρέμβασή μου. Θα συμφωνήσω ότι πριν να μιλήσουμε για την Ένωση για τη Μεσόγειο, δεν πρέπει να ξεχνάμε το ζήτημα της Παλαιστίνης και θα επανέλθω στην πρωινή μου παρέμβαση. Το ζήτημα αυτό όλοι το γνωρίζουν και ξέρουν ότι τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε, όπως ο περιορισμός της βίας, είναι στόχοι κοινοί. Ποιες όμως είναι οι διασφαλίσεις που έχουμε ότι δεσμευόμαστε να επιδιώξουμε αυτούς τους στόχους. Υπάρχουν ψηφίσματα του ΙΕ, υπάρχουν διεθνείς πρωτοβουλίες ειρήνης, υπάρχουν αμερικανικές πρωτοβουλίες προς αυτό το στόχο, όμως όλοι ξεχνούν το εξής τις αραβικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία συνθήκων ειρήνης, της σταθεροποίησης και οριστικής λύσης της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, αλλά εφόσον έχασα την ευκαιρία στην προηγούμενη συζήτηση, θα θέσω το εξή ερώτημα. Υπάρχουν ελπίδες ή έστω που μας επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε την ειρήνευση γιατί για το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και για όλους, εφόσον όλοι φαίνεται να επιθυμούν την ειρήνη, γιατί το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να επιληθεί οριστικά. Κάτι, ένα ζήτημα που πραγματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό μας απασχολεί με επεισόδια φρικαλαιοτήτων, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτιστικών δικαιωμάτων. Τι αντισταθμίσματα, τι ανταλλάγματα μπορούμε να προσφέρουμε στα θύματα για τα οποία η διεθνής κοινότητα δεν αναλαμβάνει δράση, απλώς παρατηρεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να αναλάβουν μαζί της δράση. Και έχουμε και τη συνεργασία της Βόρειας και της Νότιας Ακτής της Μεσογείου. Μιλάμε για έναν νεοσχηματιστέντα οργανισμό, ο οποίος ε, για πολλούς ακόμη δεν έχει καν δημιουργηθεί. Κάποιοι από τη χώρα με έχουν ζητήσει να τους εκπροσωπήσω εδώ. Εάν λοιπόν ε, υπάρχουν βάσεις να μην ε, έχουμε πίστη στην επιβίωση αυτού του νεογέννη οργανισμού, θα θέλαμε να το ξέρουμε, όπως και θα θέλαμε να ξέρουμε όλο αυτό το εγχείρημα τι μπορεί να μας επιτρέψει να πετύχουμε. Ίσως χρειάζεται μια νέα δομή, αλλά τι μπορούμε να διασφαλίσουμε και στους συμμετέχοντες για να αποδείξουμε την καλή μας βούληση, την καλή μας πίστη και ότι η δομή αυτή μπορεί να κρατήσει στο χρόνο και να γεννήσει λύσεις. Λύσεις για ζητήματα εκ των οποίων το σημαντικότερο είναι η συμφιλίωση και η διελεύκανση των δυσκολιών μεταξύ χωρών. Πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες και να δημιουργήσουμε την μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ περιοχών της Μεσογείου που δεν διαθέτουν και άλλων που δεν την διαθέτουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Εκτός εάν φροντίσουμε ο οργανισμός αυτός, η δομή αυτή, να λάβει υπόψη πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, το πολιτικό σκέλος και άλλα. Νομίζω λοιπόν ότι τελικά με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να είμαστε επιτυχεί στην προσπάθειά μας εφόσον οι ηγέτες και οι μας ε, ακολουθήσουν ένα ευθύ απο δράσεις Εάν όχι, δεν θα τα καταφέρουμε. Θα πρέπει όλο αυτό το ζήτημα λοιπόν να ξεκαθαριστεί. Προκειμένου να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη ένωση για την Ευρώπη, για να μην έχουμε απλώς μία πομφόλιγα σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστούμε κύριε Μπεντούμε, κύριε Σαντούκα. Έχετε ζητήσει και πάλι το λόγο. Ελπίζω θα είστε σύντομο, γιατί στην άρξη τη συζήτηση είχατε λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ε, ικανοποίησή μου για τα σχόλια κάποιων συναδέλφων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβεβαίωσαν ότι είναι αδύνατο να παραβλέψουμε το πολιτικό σκέλος της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Στο παρελθόν κάποιοι υπέθεταν ότι θα επικεντρωθούμε στο οικονομικά ζητήματα και μόνο. Όμω και οι Ευρωπαίοι συναδελφοί μου είπαν, όπω και εγώ, ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε σε καμία περίπτωση την πολιτική διάσταση. Διότι τα γεγονότα όπως ε, τα επεισόδια στη Γάζα απέδειξαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Με κάποια δυσαρέσκεια άκουσα αυτό που είπαν άλλοι, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε για πάντα μέχρι να επιληθεί η σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ή Αράβων. Διερωτώ με, γιατί κάποιοι από τους συναδέλφους πιστεύουν ότι το Παλαιστινιακό και η διένεξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων ε, θα πρέπει να διαρκεί. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν διεθνή ψηφίσματα τα οποία εάν όλοι σεβόμαστε θα έπρεπε να έχουν ήδη δώσει τέρμα στην ε, διένεξη αυτή. Δεν γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι οι χώρες που μπορούν να ασκήσουν επιρροή στον κόσμο μας, ιδίως στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες, Εάν ήταν ειλικρινείς στις προσπάθειές τους και στο πώς χειρίζονται τα διεθνή ψηφίσματα και τα άρθρα του διεθνούς δικαίου και αν δεν χρησιμοποιούσαν ε, διπλά μέτρα και σταθμά δεν γνωρίζουν ότι θα είχε επιληθεί το Μεσανατολικό και ότι οι Παλαιστίνοι θα είχαν τα πλήρη δικαιώματά τους και θα μπορούσαν να τα ασκήσουν το ζήτημα λοιπόν αυτό μπορεί να διαρκεί δεκαετίες και αυτό θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί εάν δεν δράσουμε με τρόπο ειλικρινή, έντιμο και ορθό και αν δεν φροντίσουμε για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου με ίδια συνθήκες για όλους. Θα πρέπει το διεθνές δίκαιο να μην εφαρμόζεται πλέον με τρόπο αμφιταλαντευόμενο για τους μεν και τους δε. Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι πότε ακριβώς γνωρίζουν πότε υπήρξε συνεργασία πραγματική σε επίπεδο Ευρώπης. Διότι μην ξεχνάμε τι έγινε με την ναζιστική κατοχή δεν συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά μετά. Λοιπόν, εδώ θέλουμε ισότιμες χώρες, χώρες που ισότιμα να μπορούν να συνεργαστούν. Οι Παλαιστίνοι θα πρέπει ισότιμα να συνεργάζονται με τις μεσογειακές χώρες, τις χώρες της βόρειας και της νότιας ακτής της Μεσογείου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισοτιμία. Ισοτιμία και αυτό δεν υπάρχει όταν δεν έχουμε ελευθερία μετακίνησης. Ελευθερία διέλευσης και δι... περάσματος από το ένα χωριό στο άλλο στη χώρα μας. Όταν λέμε λοιπόν κάτι, όταν κάνουμε δηλώσεις, θα πρέπει να είμαστε και συνεπίσως προς τις δηλώσεις μας. Θα πρέπει η ισοτιμία αυτή να είναι δεδομένη. Θα πρέπει η κατοχή να πάψει. Δεν μπορούμε όσο είμαστε σε κατοχή να βρισκόμαστε σε συνθήκες ισοτιμίας απαλλάξτε μας από το Ισραήλ και μετά θα μπορούσαμε να δώσουμε τα χέρια και να δράσουμε πλέον ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό μου περιγράφω ισότιμα. Όσο μας κατέχει το Ισραήλ, όσο ε, δεν έχουμε αυτή την ελευθερία, δεν μπορούμε να είμαστε ισότιμοι μαζί σας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αμπεζά από την Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σημειώσω ότι η Αίγυπτος μεριμνά ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία αυτή. Από δε την εμπειρία μας, από τις σχέσεις με τα ευρωπαϊκά κράτη, τα αραβικά κράτη, τα αφρικανικά κράτη, γνωρίζουμε ότι ο χώρος στον οποίο κινούμαστε είναι πάρα πολύ περίπλοκος, φυσικά δεν λέω τίποτε το καινούριο, έχουμε Όμω δυστυχώ μερικού οι οποίοι προσπαθούν να κοιτάξουν την Ανατολή που είναι τόσο περίπλοκη με πολύ απλοϊκέ ιδέε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει και την Ευρώπη να την αναγνωρίσουμε ω έναν χώρο αρκετά περίπλοκο από τη δική του την πλευρά και να ε, τον κρίνουμε με, τη, με τους όρους που του αρμόζουν. Όμως πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι την ιστορία την κρίνουν πολλές φορές σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική θέση ε, ξέρουμε ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη για, ως χώρος γεωγραφικός για αιώνες. Άρα ξέρουμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τον χώρο αυτό τον γεωγραφικό θα πρέπει να τον εξετάζουμε ως ένα όλο. Δεν μπορούμε την ε, συνεργασία οικονομική και άλλη να την κρίνουμε μόνο με πολιτικούς όρους. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές βέβαια στην ε, προσέγγισή μας. ε, χωρίς να ρεσμονούμε τα προβλήματα τα οποία μπορούν να τρέψουν τα πάντα ανα πάσα στιγμή στην περιοχή. Δεν μπορούμε δηλαδή ε, να μένουμε με τα χέρια δεμένα ενώπιον τέτοιων προβλημάτων. Και θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο δεδομένα. Καταρχάς ότι υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί αλλά και οι γεωγραφικοί ε, θέση που καθιστούν απαραίτητη τη συνεργασία των δύο όχθεων της Μεσογείου. Δεύτερον ότι είναι τρεις οι ήπειροι που βρέχονται από τη Μεσόγειο, τρεις ήπειροι οι οποίες έχουν δικά τους προβλήματα κάθε μια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ε, στον όρο Βόρεια Οχθή δεν ε, περιορίζονται, δεν εντάσσονται μόνο οι χώρες της Ευρώπης που βρέχονται από τη Μεσόγειο, αλλά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Όχθη της Μεσογείου ε, βρέχει χώρες που ανήκουν στην Ασιατική Ήπειρο. Έτσι λοιπόν, Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε κατά τρόπο σφαιρικό και να κοιτάξουμε τα πράγματα με τη σειρά, να μην ε, μπερδευτούμε όπως είχε γίνει στο παρελθόν στην Αίγυπτο που δεν ξέραμε αν έπρεπε να ξεκινήσουμε διαρθρωτική με οικονομική μεταρρύθμιση. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η σταθερότητα στην Μεσόγειο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εάν δεν επιληθεί το, το Παλαιστινιακό το Παλαιστινιακό, το οποίο επηρεάζει καθημερινά τη ζωή όλων των μουσουλμάνων από την Ινδονησία μέχρι τις όχθες της Αφρικής. Αυτό είναι μια προτεραιότητα. Προτεραιότητά μας είναι η πρόοδος στον τομέα αυτό και πρέπει να είναι πρόοδος στον τομέα αυτό και ελπίζουμε να μην αποδειχθεί αποτυχημένη πρωτοβουλία της Βαρκελόνης, να μην αποδειχθεί ε, αποτυχημένη αυτή η πρωτοβουλία όπως και η πρωτοβουλία της Βαρκελόνης που πέτυχε διότι είναι μόνο διμερής ε, πρωτοβουλία. Δεν μπορεί μια πρωτοβουλία αποκλειστικά διμερής να επιτύχει. Πρέπει να δούμε όλες τις διαστάσεις και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετέχουν πραγματικά στη λύση. Και μην ξεχνάμε ότι χρειάστηκε να βρεθεί μια ε, λύση, μια οργάνωση η οποία θα είναι σε θέση να συντονίσει τις δραστηριότητες και τις δύο όχθες της Μεσογείου. Σε κάθε νέα δομή όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου θα ε, ε, έχει αναμφίβολα κάποιες δυσκολίες στην αρχή, στην εκκίνησή της και μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όπως θα εμφανίζονται με τη σειρά. Δεν μπορούμε όμως να λησμονούμε τα σοβαρά ζητήματα, δεν μπορούμε να λησμονούμε τις προτεραιότητες σε ένα χώρο τόσο περίπλοκο και δεν μπορούμε παρά να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εκδηλώσουμε και την πολιτική βούληση για επίλυση των προβλημάτων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σαπουλά από την Παλαιστίνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συζήτηση είναι πολύ σημαντική σήμερα. Ανοίγει νέους διάβλους αλληλοκατανόησης Κάποιοι πιστεύουν ότι τα πολιτικά ζητήματα δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν την πρόοδο στα οικονομικά θέματα. Ωστόσο, αναμφίβολα, όλη η διαδικασία, είτε πρόκειται για τη Βαρκελόνη το 1995, από την οποία δημιουργήθηκε μετά η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και μετά η Ένωση για τη Μεσόγειο και μετά η, με, η Ένωση, η Μεσογειακή Ένωση και η Κοινοβουλευτική της Συνέλευση, Όλες αυτές λοιπόν οι διαδικασίες, οι, οι φάσεις της διαδικασίας προχώρησαν με την προοπτική ότι προχωρεί προς επίλυση μια σειρά διενέξεων της περιοχής και ότι έτσι χρειάζεται οργάνωση για να προχωρήσουμε περισσότερο. Με την αίσθηση ότι είμαστε ε, όλοι ε, κοινωνοί της ίδιας ιστορίας, της ίδιας γεωγραφίας, έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Ασφαλώς και η σταθερότητα ή αντίστροφα η κρίση, η σύγκρουση σε οποιαδήποτε περιοχή, σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής μας, του χώρου μας, του γεωγραφικού, θα επηρεάσει κάποιο άλλο ε, σημείο. Εμείς Παλαιστίνοι λοιπόν είμαστε μέλος αυτής της διαδικασίας, μέλος της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Υπάρχει άλλη χώρα όμως η οποία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα που που διαπράττει εγκλήματα που όπως είπε και ο ίδιος ο δικαστής Goldstone στην έκθεσή του θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να παραμείνουμε σιωπηλοί ότι είμαστε θύματα τέτοιου είδους αδικίας ή ότι θα έπρεπε οι άλλοι να παραμένουν σιωπηροί ε, και να παρακολουθούν αμέτωχοι τη διεξαγωγή αυτών των σφαλμάτων, αυτών των αδικημάτων, αυτών των εγκλημάτων. Ε, ερωτώ, όταν στην Αυστρία θεωρήθηκε ένα κόμμα πως, ε, το οποίο είχε ψηφιστεί ότι δεν ακολουθεί τις αρχές, ε, την, ε, το πολιτικό σορθόν, τα παραδεδεγμένα της δημοκρατίας. Πώς αντέδρασε η Ευρώπη το αυτό κόμμα εξελέγει. Δεν την έβαλε την Αυστρία ολόκληρο στο περιθώριο. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι μας αντιμετωπίζουν με ισότιμους όρους, με ίσα μέτρα και σταθμά. Όπω είπε και ο σα, πρέπει να είμαστε θέση να κοιτάξουμε ο στον τον άλλον στα μάτια με σεβασμό, σε βάση ισότιμη. Πώ λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε αν αυτό δεν είναι δυνατόν. Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμεθα την, εγκληματικέ τις εγκληματικές ενέργειες, τις διακρίσεις μα. βάρος μας, ε, πρακτικές οι οποίες προσωμιάζουν στο Απαρτχάιτ, Πώς λοιπόν είναι δυνατόν εμεί ή οποιαδήποτε χώρα να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και να ε, κοιμούμαστε ήσυχοι το βράδυ. Όταν μιλούμε για συνεργασία, συνεργασία σε κάθε τομέα, ναι, συνεργασία και σε επίπεδο ανθρώπινο, χωρίς ιδιωτελή συμφέροντα. Έστω και αν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέσεις μεταξύ κρατών που να μην στηρίζονται στα αμοιβαία ιδιωτελή συμφέροντα, που να μην στηρίζονται σε ένα κοινό παρανομαστή που να μας ενώνει, που να μας φέρνει πιο κοντά. Εάν λοιπόν δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε η μεν τις ανάγκες των δε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε κατά τρόπο ενωμένο, ενωτικό, σε συνεργασία και σεβασμό αμοιβαίο. Και ως εκ τούτου, εμείς Παλαιστινοί, δεν θέλουμε να χρονοτριβούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα περιμένει για να προχωρήσουμε στη συνεργασία. Ένα παράδειγμα, εδώ σήμερα το πρωί, όταν όλοι κατεδίκασαν το Ισραήλ, τις πρακτικές του, την ε, ε στρατιωτική επίθεση εις βάρος της Γάζας. Από χώρες που δεν είχαν άμεση εμπλοκή με την ε, Παλαιστίνη ή τα, τα αιτήματα των Παλαιστινίων. Και από την άλλη ακούμε ότι πρόκειται να υπογραφεί συμφωνία άνευ προηγουμένου με το Ισραήλ. Πώς είναι δυνατόν το Ισραήλ να αντιληφθεί ότι η κατοχή εδαφών άλλης χώρας, ή άδικες και παράνομες με βάση το διεθνή δίκαιο επιθέσει του στρατιωτικέ επιθέσει δεν θα έχουν επιπτώσει, εάν από την άλλη πλευρά ε, του ανοίγουμε αγκάλες και το υποδεχόμαστε στους κόλπους μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν λοιπόν πρόκειται να προχωρήσουμε ουσιαστικά και πραγματικά, θα πρέπει να μιλούμε όχι μόνο για το ίδιο τελέσμα συμφέρον ο καθένας, αλλά να σεβόμεθα και το συμφέρον του άλλου. Μόνο έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε ένα τον άλλον. Εάν πείσουμε, εάν δείξουμε στον εγκληματία ότι πρέπει να πληρώσει το τίμημα του εγκλήματός του, όπως τον Κόλστον την προηγούμενη εβδομάδα στην Νέα Υόρκη με την έκθεσή του, που είπε ότι αυτό είναι και το νόημα της έκθεσης. Δεν θα κερδίσει τον πόλεμο, δεν θα φέρει την λύση στην ε, ε Μέση Ανατολή, αλλά θα δείξει ότι ο εγκληματίας τιμωρείται για το έγκλημά του. Ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και ότι καμία χώρα δεν βρίσκεται στο απειρόβλητο των αδικημάτων, που, των συνεπειών μάλλον των αδικημάτων που διέπραξε. Εάν λοιπόν πρόκειται να συνεργαστούμε, θα πρέπει να δούμε και κάποια θετικά μηνύματα που θα μας φέρουν πιο κοντά. Η παράδοσή μας, οι πολιτιστικές μας ρίζες, μπορεί να λένε πρέπει να μπορεί να λένε στηρίξτε κάποιον ακόμη και αν έχει άδικο. Στηρίξω το φίλο σου ακόμη και αν έχει άδικο. Είναι δυνατό να μου στέλνετε κάτι τέτοιο. Θα το στηρίξω και όταν έχει άδικο. Παρα... Με... Ο μόνος τρόπος να στηρίξει τον έχει άδικο είναι να του πω ξεκάθαρα, κοίταξε έχει κάνει κάτι λάθο, έχει άδικο, διορθωσέ το. Μόνο έτσι μπορώ να τον στηρίξω και να είμαι πραγματικό του φίλο. Εάν ακολουθήσουμε λοιπόν μια τέτοια πρακτική, πιστεύω μπορούμε να προσεγγίσουμε μεν του δε. έτσι ώστε το εγχείρημα στο οποίο αποδιόμαστε να στεφθεί με επιτυχία και να μην ε, αποτύχει παταγωδός όπως τα προηγούμενα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε τον επόμενο Γενάρη να έχουμε ένα φύλλο πορείας, αλλά πείτε, επιτρέψτε μου να πω, ένα φύλλο πορείας που θα ορίσει όρους κατάλληλους να περιοριστούν οι εγκληματικές ενέργειες, τα δεινά και να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η ελευθερία στην περιοχή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέλα από τη Μάλτα παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. In my opinion, <clears throat> started on a very good footing. The idea of Sarkozy was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 θα πρέπει να δείξουμε ανοχή ε. στις, ε, στις πεπιθήσεις σημαίνει των Να βρούμε σημεία σύγκλησης και σημεία απόκλησης μεταξύ ημών και εταίρων. Δυστυχώς, Project. Θεωρούν αυτή την υπόθεση σαν μια υπόθεση ε, ευρωπαϊκή. Είναι κάτι δηλαδή που ξεκινάει από την Ευρώπη και πηγαίνει προς τον Νότο. Είναι ε, ένα φετφά που επιβάλλεται από τον Βορρά στον Νότο. Ε, δηλαδή ότι προσπαθούμε να του επιβάλλουμε τι αξίε τι ε, ευρωπαϊκέ στις, κουλτούρε, στου στους πολιτισμούς της Βόρειας ε, Αφρικής. Ακόμα και η δημοκρατία, ακόμα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μα τι, ενώ πώ συλλαμβάνουμε την έννοια τη δημοκρατία. Τι βασικέ έννοιε. Άλλα εννοούμε στην Ευρώπη περί αυτό και άλλα στην Βόρεια Αφρική. Επομένω, θα πρέπει να δούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλιώ θα έχουμε κάθε αξιοπιστία. Τώρα, όσον αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση, είναι κάτι πολύ βασικό. Αυτή τη 14 ετία, από το 1995 και μετά, τι καταφέραμε ε, όσον αφορά τον αναλφαβητισμό στι ε, χώρε εκείνε. Ε, η διακίνηση των φοιτητών των σπαστών έγινε πιο εύκολη, ήρθαν κάποιοι περιορισμοί θεωρήσεων διαβατηρίων. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κάτσουμε και να ξεκινήσουμε από το α. Από τη βάση, από τα θεμέλια και όχι από το διακυβερνητικό επίπεδο να κατέβουμε προς τα κάτω. Και θα πρέπει ομένως να κάτσουμε και να οργανώσουμε, να γίνουμε sponsors, χορηγοί σε κάποιες εκδηλώσεις πολιτικές και έτσι να μπορεί ο κόσμος να συνευρεθεί γύρω αυτές τις πολιτικές εκδηλώσεις γιατί κάτσαμε και τους ε, μιλήσαμε για μια ευρωμεσογειακή ε, ένωση ελευθερών εμπορίου. Έγινε τίποτα. Υποτίθεται ότι από του χρόνου θα, θα, θα, θα αρχίσει να τρέχει. Όχι. Ε, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα για πλευρά των αραβικών χωρών. Από την άλλη μεριά όμω είναι, είναι πάρα, πάρα πολύ μικρέ, πάρα πολύ λυπή και ανεπαρκεί οι επενδύσει οι ευρωπαϊκέ στι χώρε εκείνε. Να, μερικά από τα ζητήματα που μπορούμε να επισημάνουμε, κυρία Πρόεδρε. Ε, και, και προσπαθώ να είμαι σύντομο γιατί ξέρω ότι πιέζει ο χρόνο. Όμω πριν φτάσουμε στα πιο σημαντικά πολιτικά ζητήματα, αυτά που θα πρέπει εδώ να τα επιλύσουμε, θα πρέπει πρώτα να πω σε αυτέ τι μεταβλητέ, όπω είπα, την, ε, την παιδεία, τι διαπολιτισμικέ σχέσει ε, και τη θρησκεία. Όλα αυτά για, για, για, για τι δύο χθε του Μεσόγειου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κύριε Βέλλα, ευχαριστώ πολύ πρώτο και τώρα δώσουμε τη σκητάλη στον κύριο Χασντάουι που προέρχεται από την Ιορδανία. ευχαριστώ, κύριε Ραΐς. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε... Θα ήθελα να θίξω κάποια ζητήματα για να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε σε σχέση με την ε, ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση. Θα επιστρέψω στο 1993 όταν εργαζόμουν στο στρατό και ο κύριος Χουσέν μας ε, επισκέφθηκε και μας μίλησε για τις επιλογές της Μέσης Ανατολής. Μια από αυτές τις επιλογές ήταν η ειρήνη. Από τότε μιλάμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Όμως φαίνεται ότι αυτό παρέμεινε μια ελπίδα φρούδα που ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα. εάν έχουμε δαπανίσει όλα τα κονδύλια που διαθέταμε για όπλα, για πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Εάν τα είχαμε δώσει για την παιδεία και τον πολιτισμό, ίσως να είχαμε πετύχει πολύ περισσότερα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι υποσχέσεις δεν μπόρεσαν να γίνουν πράξη και δεν εμποδίσαμε τα παιδιά μας να κοιτάζουν στην τηλεόραση τους φόνους και τις δολοφονίες που έγιναν. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε τα παιδιά μας να μην βλέπουν πλέον τέτοιες σκηνέ. Έστω και στι οθόνε τη τηλεόραση. Θα πρέπει να τα γαλουχίσουμε με τι αρχέ τη ειρήνη. Άκουσα τον ε, πρόσωπο του Ισραήλ, ο οποίο μίλησε και ε, ελπίζω ότι αυτό θα γίνει για την αποχώρηση του Ισραήλ από την Γάζα. Ακούσαμε το τι συζητιέται και τι συμβαίνει με την ε, με τον ελιμενισμό πλοίων στην ε, Γάζα, με, τον, ε, με, τη, με τα αεροδρόμια. Φαίνεται ότι όλα αυτά όμως παραμένουν όνειρα. Εγώ το προηγούμενο όνειρό μου το είχα βασίσει στην ελπίδα. Τώρα φαίνεται ότι βρίσκομαι πια στο επίπεδο της φαντασίωσης. Δεν έχω ελπίδες όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Άκουσα και τους συναδέλφους από το Ευρωκοινοβούλιο και παρατηρώ ότι πολλοί πιστεύουν ότι η ενίσχυση των οικονομιών μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία ειρήνευσης. Πώς όμως μπορούν να ανθρωπιοποιήσουν σε συνθήκες κατοχής μέσω οικονομικής μεταρρύθμισης να βελτιώσουν τι σχέσει του με του κατακτητές του, τι οικονομικέ δραστηριότητε να αναπτύξουν. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν απελευθερωθούν. Μην ξεχνάμε τι έγινε στην Νότια Αφρική. Εκεί όλες οι χώρες κατήγγυλαν το Απαρτχάιτ και μόνον όταν ο αφρικανικός λαός ε, κατέκτησε την ελευθερία του μπόρεσε να αναπτυχθεί και οικονομικά. Ή το καθεστώς στο Ιράκ. Όταν θεωρήσαμε ότι το καθεστώς αυτό ήταν παράνομο, τότε είχαμε τη διεθνή παρέμβαση. Οι διεθνείς δυνάμεις προσπάθησαν να επιβάλλουν τα ψηφίσματα για τι αποφάσει του ΟΗΕ. Όμω αυτό δεν συμβαίνει για την ώρα στην Παλαιστίνη. Το Ισραήλ δεν εξαναγκάζεται να εφαρμόσει τι αρχέ του διεθνού δικαίου. Στο κράτο αυτό λοιπόν της Παλαιστίνης, τι σχέσεις εταιρικέ και οικονομικές να αναπτυχθούν με άλλες χώρες. Εάν το ζήτημα αυτό επιληθεί, ναι, η οικονομία μπορεί να λάβει και πάλι τη σημασία που τη αξίζει. Όμως αυτό δεν θα γίνει υπό συνθήκες κατοχής. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να θυμίσω αυτό που είπε και ο κύριος Σαρκοζή, ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι ένα μεγάλο όνειρο. Και όπως είπε και ο κύριος Χουσίν, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δρόμος για να γίνουν τα όνειρα πράξη μπορούν να περνούν μόνο μέσα από τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Ειρήνη για όλους τις περιοχές μας. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Χαουάστει. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κάλσον, ο οποίο θα επιχειρήσει να απαντήσει σε ορισμένε από τι ερωτήσει που του τέθηκαν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μορένο, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου, για μια σύντομη παρέμβαση και για να έχουμε και την άποψη τη κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Είμαι σύντομο. Θα πρέπει να κάνετε και να λάβετε υπόψη το τι έγινε όσον αφορά αυτή την διακήρυξη ε, του, Συμβουλίου, Οικονομικών και Γενικών Θεμάτων που έγινε στην Αλεξάνδρεια ε, διότι θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι σε εκείνη την ετησία συνάντηση η οποία έλαβε χώρα με την συνεργασία ε, του οργανισμού, του μη κυβερνικών οργανώσεων, της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και διάφορων οικηφορείων της Αιγύπτου. Ε, συζητήθηκαν τα ζητήματα τα σχετικά με την ειρήνη, με την έλλειψη της ειρήνης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, ούτω ώστε οποιαδήποτε θεματική να αναστέκει. Ε, γιατί έχουμε πάρα πολύ συμβατικά πράγματα, ζητήματα όπως την, την ανεργία, την μετανάστευση και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να, αντιμετωπίσουμε ούτω ώστε να δούμε ποιο θα είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών υπομορφή δομημένη, οργανωμένη ε, στα πλαίσια της ε, Μεσογείου και ε, γίνανε κάποια βήματα πρόοδου ώστε έχουμε αυτό το, το δίκτυο των οικονομικών και κοινωνικών συμβουλίων, ούτω ώστε αυτή τη στιγμή για να μπορεί να υπάρχει ένα ένας διάλογος που αν θεωρήσουμε ότι θετική εξέλιξη επίση. Ε, τρία ήταν τα θέματα που θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να μελετηθούν, να ζητηθούν μέχρι την επομένη ετησία τέτοια ε, συνάντηση. Και θα να σας τα πω ποια θα είναι ε, σύντομα. Πρώτα πρώτα, να δούμε πώ μπορούμε να δουλέψουμε όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, να δούμε πώ θα πετύχουν περισσότερη απασχόληση και ανταγωνιστικότητα. Δεύτερον, να υπάρχουν αξιοπρεπεί όροι εργασία ε, σχετικά με τα, με, θέματα του, του μου, του συνεταιρίζεστε και αυτά. Και επίση θα πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και να αποπτέσουμε το τι γίνεται όσον αφορά το τι θα κάνουμε για να κατοχυρώσουμε, να βαθύνουμε το ρόλο τη γυναίκα στην κοινωνία. Euh, Ευχαριστώ κύριε Μορενό. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κάλσον για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις απαντήσεις μου. Ομαδοποιώντας τις ερωτήσεις. Όσον αφορά τις σχέσεις ε, της Ένωσης για τη Μεσόγειο και την ε, διαδικασία για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Ήταν σαφές νομίζω σήμερα το πρωί που ήταν ε, στη θέση μου εδώ καθισμένος ο συνάδελφος και προϊστάμενος μου ότι προφανώς εμπλέκεται στη διαδικασία για την ειρήνευση η Ένωση για τη Μεσόγειο. Επίσης Η Ένωση για τη Μεσόγειο πρέπει να πούμε βεβαίω ότι δεν αποσκοπεί στην επίλυση τη λύση. Μεν. Πλην όμω, όπω και η διαδικασία τη Βαρκελόνη προηγουμένω, έχει αποδείξει ότι δεν ε, λειτουργεί εν πολιτικό κενό και ότι δεν μπορεί παρά να συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ως εκ τούτου να ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή, η επίλυση της διαφοράς. Ξέρουμε βεβαίως ποια είναι τα προσκόμματα που μπορεί να προξενεί μια τέτοια σύγκρουση στην πολυμερή συνεργασία. Πιστεύουμε ωστόσο ότι η Ρώση και τη Μεσόγειο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για επικοδομητικό διάλογο δεδομένου ότι 43 εταίροι, μεταξύ των οποίων και οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση, βρίσκονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Επίσης προσφέρει και ένα εργαλείο χρήσιμο πιστεύουμε, αν όχι άμεσα πάντως μακροπρόθεσμα, είναι φθέτο χρόνο και όταν υπάρχουν καλύτερε προοπτικέ, η Ένωση για τη Μεσόγειο. Μπορεί να αποτελέσει λοιπόν ένα χρήσιμο εργαλείο, όπω είπατε και κάποιοι από εσά, όντω είναι ένα μακροχρόνιο, μακροπρόθεσμο εγχείρημα. Και Ω προ τη σύγκριση, μετα... τη σύγκριση μεταξύ διαδικασία Βαρκελόνη και Ένωση για τη Μεσόγειο, ναι, θα μπορούσε να αποτελέσει η Ένωση για τη Μεσόγειο ένα μεταγενέστερο στάδιο, αν θέλετε. Δηλαδή, στηρίζεται πάνω στη Βαρκελόνη και θα ήταν εσφαλμένο το να θεωρήσει κανεί ότι ανήκει μόνο στο παρελθόν ε, είναι κομμάτι μόνο της ιστορίας η διαδικασία της Βαρκελόνης. Ε, μπορεί μόνο πάνω στη Βαρκελόνη στηριζόμενη να αποτελέσει επιτυχή ε, προσπάθεια η Ένωση για τη Μεσόγειο. Ωστόσο θα πρέπει ταυτόχρονα να δοθεί και έμφαση σε συγκεκριμένα σχέδια, λαμβανομένων υπόψη ε, και των 13 ετών εμπειρία που έχει να προσφέρει η διαδικασία της Βαρκελόνη, η οποία με την διατομεακή της προσέγγιση, ασφάλεια, οικονομία και διαπροσωπικές ε, σχέσεις, οι διανθρώπινες σχέσεις, μπόρεσε να προχωρήσει σε όλη αυτή την περίοδο. Η μετάβαση μεταξύ Ευρωμεσογειακής και Ένωσης για τη Μεσόγειο ε, μπορεί να γίνει με τη διατήρηση συμπροεδρίας, με μία μόνιμη επιτροπή, με μία μόνιμη γραμματεία που θα εδρεύει στη Βαρκελόνη και που θα παρακολουθεί τους έξι τομείς ε, πολιτικής που ενέκρινε η διάσκεψη των Παρισίων. Χτυπάει το, το τηλέφωνο του ομιλητή δυστυχώς. Πολλά ήταν τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν ως προς την γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ και σε αυτά. Καταρχάς, Όπως είπα στην αρχική μου παρέμβαση, ο Γενικός Γραμματέας θα προέρχεται από ένα από τα ε, κάθε της Μεσογείου. Όταν μιλούμε για αναπληρωτές γενικούς γραμματέης ε, που ανέφεραν ε, στα παραδείγματα τους κάποιοι από τους ομιλητές, ίσως να γνωρίζετε ήδη, ότι για την πρώτη τριετία τις θέσεις αυτές έχει προβλεφθεί να καταλάβουν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, και ελπίζουμε να καταλήξουμε συμφωνία και για την έκτη θέση αναπληρωτή από την Τουρκία. Η Συμπροεδρία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις ως προς το θέμα των αναπληρωτών γενικών γραμματέων. Ασυστά ακόμη και τον αριθμό των θέσεων γενικών γραμματέων, αλλά και τα χαρτοφυλάκια που θα αναλάβουν. και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε κάποια λύση μέχρι τα τέλη του μήνα. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσω για τη γραμματεία ότι θα, επικεντρωθούμε σε, θα επικεντρώνεται μάλλον σε σχέδια, project και θα έχει τεχνικό χαρακτήρα. Τα project θα ακολουθούν τις προτεραιότητες όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο Παρίσι και τη Μασαλία. Δηλαδή ρήπανση, ενέργεια, εκπαίδευση, μεταφορές, οικονομική ανάπτυξη, προστασία των πολιτών, πολιτική προστασία. Θα επεκταθώ λίγο περισσότερο στα, στα project αυτά, ναι, και το ζήτημα. Υπάρχουν ιδέες που έχουν προβληθεί για όλους τους τομείς. Κάποιοι από τους εταίρους έχουν αρχίσει συζητήσεις. Κάποιες προτάσεις ήδη έχουν ε, προχωρήσει. Για δε τη χρηματοδότηση πολλοί διεθνεί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπω Διεθνέ Χρηματοπιστωτικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρω... Αραβική Τράπεζα Επενδύσεων, μάλλον Ευρωπαϊκή Τράπεζα, συγγνώμη, Αραβική Τράπεζα Ανάπτυξη, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Χρηματοδότηση επίση θα προέλθει και από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχει προσημειωθεί το ποσό που αφορά την ε, Μεσόγειο ε, και βέβαια θα υπάρξουν και ε, χορηγίες, τελωτικές δηλαδή εισφορές. Θα υπάρξει επίσης υποστήριξη από ειδικού προερχόμενους από τα κράτη-μέλη. Σημαντικό όμω είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε την σύσταση της ε, ε, γραμματείας. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εξασφάλιση στη χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση. Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα τα οποία καθιστούν τόσο σημαντική την εξέβρεση λύσεως προς το καθεστώς. Γι' αυτό καταβάλουμε τόσο σημαντικές προσπάθειες. Έχουμε αρχίσει επίσης να ε, λαμβάνουμε, να παραλαμβάνουμε συγκεκριμένα project, όπως είπα, σχέδια, ε, Όμω δεν μπορούμε να του δώσουμε συνέχεια όσο δεν έχει επιληθεί το ζήτημα τη γραμματεία και όπω είπα και στην προηγούμενη μου παρέμβαση, ελπίζουμε στι αρχέ του προσεχού έτου να έχουμε κατάληξη. Ε, Πάντω, όλε μα οι προσπάθειε ε, κατευθύνονται προ το αυτό. Θα στραφώ τώρα σε κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Ναι, θα μπορούσα ακόμη να επεκταθώ προς τα project ότι έχουμε παραλάβει πάνω από 30 προτάσεις. Όπως είπα όμως θα τα χειριστεί όταν έρθει η ώρα η γραμματεία. Και το ίδιο ισχύει και για την χρηματοδότηση. όσον αφορά την σημασία του διαλόγου μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών παραδόσεων και θρησκειών της περιοχής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την ύπαρξη του θεσμού που αναφέρθηκα και στον οποίο αναφέρθηκα και νωρίτερα, αλλά το Ίδρυμα Άννα Λίντ, που στόχο έχει να διευκολύνει και να προωθήσει το διάλογο, να προαγάγει το διάλογο μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων. Εδρεύει στην Αλεξάνδρεια, στην Βόρεια και έχει παρουσία και ε, Αιγυπτιακών και Σουηδικών ε, Ιδρυμάτων. Στη σύστασή του έχει δε ως Ίδρυμα δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στον διάπολιτισμικό διάλογο. για το ελεύθερο εμπόριο. Είναι πολύ σημαντικό και το ελεύθερο εμπόριο ασφαλώ. Ίσως το 2010 να είναι υπερβολικά αισιόδοξο στόχος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη ενός ε, χώρου ελεύθερου εμπορίου ε, το ταχύτερο δυνατό. Έτσι λοιπόν με τη συνάντηση στις 9 Δεκεμβρίου των ε, Υπουργών Εμπορίου εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, μπορούμε να ελπίζουμε κάποια πρόοδο, εξελίξεις ή επιτυχία ίσως έτσι ώστε να ολοκληρωθεί μια ακόμη φάση προς την ολοκλήρωση ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών. Τώρα θα προχωρήσω σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ε, ανθρώπινα δικαιώματα αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, ε, ετέθη το ζήτημα και νωρίτερα σε κάποια παρέμβαση, είναι όπως γνωρίζετε κάτι το οποίο αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση προτεραιότητα και συζητείται και στα Συμβούλια Σύνδεσης αλλά και σε διμερές επίπεδο. Και με αυτά πιστεύω, ελπίζω να κάλυψα στο μεγαλύτερο μέρος τους στις ερωτήσεις. Ο κύριος Σαντούκα θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση στον κύριο Κάλσον, ερώτηση. Θέλετε να να κάνετε τοποθέτηση μόνο ή ερώτηση. Παρέμβαση. Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση. Μπορώ να λάβω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα για την ελευθερία έκφρασης και την ανοίξη θρησκεία κοιτάξτε, δεν θα ξανανοίξουμε τη συζήτηση λέει πρόεδρο. Βάλτε τα ακουστικά σας αν θέλετε. Δεν θα ξανανοίξουμε τη συζήτηση, διότι παρεμβήκατε δύο φορές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Κάλσον απάντησε στον γύρο παρεμβάσεων Υπάρχουν ε, μέλη που δεν παρενέβησαν καν. Θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Κάλσον ή να κάνετε μια νέα παρέμβαση. Δεν είχατε διερμηνία. Θα ήθελα, ήθελα να τοποθετηθώ. Όχι να γύρω το θέμα της θρησκείας και της ελευθερίας έκφρασης ακριβώ, αλλά επειδή έχω μια συγκεκριμένη άποψη για το θέμα αυτό, ήθελα να την αναπτύξω, εάν έχουμε τη δυνατότητα. Πρόκειται για ένα νέο θέμα, άλλωστε. Η θρησκεία είναι κάτι που δεν συζητήθηκε προηγουμένω. Και μια άλλη πτυχή, η ελευθερία τη έκφραση. Δεν είναι κάτι που το αναπτύξαμε. Ήθελα λοιπόν τη δυνατότητα να τοποθετηθώ προ αυτό. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε υπό το σημείο 7, κύριε Σανδούκα, για να τοποθετηθείτε, εντάξει. Ωραία, πολύ ωραία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Κράτσα η ε, κυρία Γκράτσα ήρθε με κάποια καθυστέρηση στο μέσο συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, λυπάμαι και εγώ για την καθυστέρηση, αλλά ξέρετε γίνονται παράλληλε εργασίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να είμαι στην Επιτροπή Περιφερειακής πολιτική. Ε, ήθελα καταρχά, καταρχάς, ε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, δεν ξέρω αν το συζητήσατε, ε, να απευθυνθώ στον κύριο Κάρσον, να ρωτήσω αν προβλέπεται να γίνει η διπουργική ε, Υπουργών Εξωτερικών ε, Υποθέσεων της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, η διάσκεψη η οποία ήταν να γίνει στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο. και επίσης ήθελα να ρωτήσω εάν ασχοληθήκατε καθόλου να σχολιάσετε το θέμα των προεδρικών εκλογών πώς ε, εξελίσσεται στην ε, Παλαιστίνη, είναι άμεσα συνδεδεμένο και με την, ε, το ρόλο του Προέδρου Αμπούντα και με τις επιπτώσεις που έχει η, εμπλοκή στις συνδυνευτικές διαδικασίες στο δικό του image και στο δικό του βάρος στο πολιτικό και στη σχέση του με, την, με τη Χαμάς και την κατάσταση στη Γάζα και ε, επιπλέον επιτρέψτε μου να ε, κάνω μια διευκρίνηση όσο δεν κατάλαβα εγώ καλά για το Ίδρυμα Άννα το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό Ίδρυμα και το υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν μετέχουν μόνο εκπρόσωποι από την Αίγυπτο και από τη Σουηδία αλλά από όλα τα κράτη της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Είναι μια πληροφορία, επιτρέψτε μου να τη δώσω, επειδή εγώ άκουσα στη μετάφραση ότι μετέχουν μόνο από τη Σουηδία και από την Αίγυπτο Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πληροφόρηση για όσους δεν την έχουν, ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει μια αντένα του Ιδρύματος Αναλύν, την οποία μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και σε επίπεδο εθνικό, αλλά και σε επίπεδο διακρατικό. Κύριε Κάλσον. Θα ήθελα καταρχάς να στήσω συγγνώμη που δεν ήμουν σαφής. Ναι, βεβαίω το Ίδρυμα είναι ε, Ίδρυμα της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Δεν υπάρχει εμβολία και γι' αυτό ακριβώς και το παρουσίασε ως υπόδειγμα, ως παράδειγμα των ε, επιτευγμάτων μας και της διαπολιτισμικού διαλόγου των διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν που δεν ήμουν σαφής. Είχατε απόλυτο δίκαιο. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε για την αναβολή της ε, υπουργική στις Κωνσταντινούπολος. Μάλιστα. Όπως γνωρίζετε, είχε αρχικά προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις 24 και 25 Νοεμβρίου εφέτος. και λόγω των πολιτικών δεδομένων, των πολιτικών συνθήκων, πιστώσαμε ότι δεν ήταν δυνατό να διοργανωθεί, να διεξαχθεί τώρα ακριβώς. Αναβάλλεται, δεν ματαιώνεται και εξετάζουμε ακόμη, μελετούμε ακόμη τον τρόπο να προγραμματίσουμε να προετοιμαστεί αυτή η υπουργική διάσκεψη, λέει, το πρόγραμμα που θα πρέπει να υιοθετηθεί. και την ε, έγκριση του προγράμματος από τους αξιωματούχους του προγράμματος της ε, Υπουργικής. Επίσης, στο καθεστώς της γραμματείας, στο οποίο αναφέρθηκα, την εκλογή του Γενικού Γραμματέα και όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα έπρεπε να απασχολήσουν την Υπουργική Διάσκεψη, αλλά ε, δεν έχουμε αφήσει κατά μέρος. Τα προωθούμε και αυτά, όπως ελπίζω να εξήγησα σήμερα, γιατί τα θεωρούμε σημαντικά. Έχουν ύψιστη σημασία για την επιτυχία την ίδια της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Στόχος μας, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, αλλά και πέραν αυτής, ως τμήμα μιας συνένεσης, θα ήταν το ταχύτερο δυνατό, μόλις δηλαδή το επιτρέψουν οι συνθήκες, να διεξαχθεί η Υπουργική Διάσκεψη Ας δούμε όμως πρώτα τα πολιτικά ζητήματα και ας, δούμε, και ας αφήσουμε για μετά το χρόνο-διάγραμμα, Δηλαδή το διάγραμμα θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη ευνοϊκών συνθήκων και όρων. Ευχαριστώ και ελπίζω να είναι ικανοποιητική η απάντησή μου. Ευχαριστούμε κύριε Κάλσον. Ευθύ αμέσω να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Σα ευχαριστώ για την ε, παρουσία σα εδώ. Ξέρω ότι πρέπει να προλάβετε μια πτήση. Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε τώρα τη συζήτηση και θα περάσουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξη. Ευχαριστώ κύριε Κάρλσον. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 7. 7. Ε, μια ειδοποίηση, Πρόεδρε, πριν περάσουμε στο σημείο 7. για την Ένωση για τη Μεσόγειο, αυτό το μεγάλο εγχείρημα, να πω το εξή, ένα μήνυμα προς την συνέλευσή μας. Η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι ένας τίτλος πολύ ευρύς. Πώς μπορεί να υπάρξει πολιτική, πολιτικό νόημα εδώ. Εγώ για να έρθω σε αυτή τη συνάντηση υπέβαλα αίτηση για θεώρηση πριν από 15 μέρες. Η αντιπροσωπεία της χώρας μου υπέστη σωματικό έλεγχο. Μας πήραν και δακτυλικά αποτυπώματα. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος ε, μετάβαση δεν είναι εξωπρεπής. Πού είναι η Ένωση για τη Μεσόγειο. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να μου πείτε ότι αυτό δεν βρίσκεται στην ημερησία διαταξή σημείο, αλλά δράση πρέπει να αναλυφθεί για να έχουμε μια θετική συνεργασία μεταξύ Βορρά και Νότου. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Εγώ έχω εργαστεί ως πρέσβης της χώρας μου και σε κάθε μια από τις πρεσβείες όπου εργάστηκα ε, η θεώρηση αποστέλλεται διαλληλογραφία σε όσους τη ζητήσουν. Θέλουμε λοιπόν παρόμοιες διαδικασίες, ε, ίση μεταχείριση. Θέλω να καταγραφεί τουλάχιστον στα πρακτικά για την ερχόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Κύριε Ντάντ, σας ε, έκαναν σωματικό έλεγχο πού? Στο αεροδρόμιο? Μάλιστα. Όχι, πρόεδρε, στην πρεσβεία, στη γερμανική πρεσβεία, όταν επέβαλα αίτηση για τη θεώρηση. Διότι η γερμανική πρεσβεία είναι υπεύθυνη για την εκχώρηση θεώρησης εμάς. Σα έκαναν σωματικό έλεγχο σε πρεσβεία. Σε πρεσβεία. Ναι, μου κάνανε σωματικό έλεγχο στην πρεσβεία. Στη Δαμασκό, η γερμανική πρεσβεία, σας κάνει σωματικό έλεγχο. Πήγατε να κάνετε αίτηση για θεώρηση διαβατηρίου και σας κάνανε σωματικό έλεγχο. Υπάρχει Γερμανός ε, συνάδελφος εδώ, υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Παράξενο μου φαίνεται. να σας απαντήσω. Και η Βελγική, η Βελγική μάλλον πρεσβεία μας έστειλε, μας παρέπεμψε στη Γερμανική πρεσβεία. Διότι εκεί υπάρχει το, ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα. Και με αυτά έγινε έλεγχος, επιθεώρηση σε όλα τα μέλη της Συριανής, Συριανής αντιπροσωπείας. Κύριε Χάντατ, μήπως ήταν απλώς θέμα ασφαλείας κατά την είσοδο μέσα σε ένα Εκτός και αν ο κύριος Ράιντελ θέλει να μας πει δύο λόγια γι' αυτό. Όχι. Κοιτάξτε, υπάρχουν όροι διεθνείς για το πώς μπαίνει κανείς με βάση το στη συνθήκη του Σέγγεν επί παραδείγματι πρέπει να γίνεται ένα έλεγχο ασφαλεία ενδεχομένω ότι χρειάζεται ιδιομετρική εικόνα. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται για τα διαβατήρια όλων ημών στο χώρο του Σέγγεν δεν μπορεί κανείς να πάρει διαβατήριο αν δεν έχει τη βιομετρική εικόνα. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό διαδεδομένο. Η Πρόεδρος. Καλώς, προχωρώ στο σημείο 7 της ημερησίας διατάξεως. Πριν όμως από αυτό, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντελπίκα, ο οποίος ύστερα από τα όσα μας είπε το πρωί, θα κάνει πρόταση διακήρυξης της Επιτροπής. Πολύ γρήγορα όμως, γιατί και ο κύριος Οβιόλ ξέρω ότι βιάζεται να λάβει το λόγο. Όχι, όχι, 30 δευτερόλεπτα μόνο, Γομπέρντελ Πικά. Αν συμφωνήσετε θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την διακήρυξη για την Επιτροπή. Ναι, διότι θα υπάρξει μια δήλωση, μια έκθεση μάλλον της ε, ε, συνεδρίασης, που αφορά τη συνεδρίαση και για την επόμενη ε, συνεδρίαση. Όχι τώρα το απόγευμα, αλλά σήμερα το πρωί θα θυμάστε ότι προ το τέλο τη ε, συνεδρίαση έλαβα το λόγο για να πω ότι πρέπει να ληφθούν όλα όσα είπαν οι μεν και οι δε, αλλά κατά τρόπο απλό, χωρί να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα περίπλοκο που θα περιπλέξει τα πράγματα και θα μα ξαναρίξει στις, ε, στα ιωθώτα. Γι' αυτό λοιπόν και αν δεν κάνω λάθο, ο συνάδελφο από την Αίγυπτο είπε κάτι αντίστοιχο, ο κύριο Λεμπίτ, ότι δηλαδή θα πρέπει να αποφύγουμε τα μεγάλα ψηφίσματα. Αλλά από την άλλη πρέπει κάτι να δηλώσει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης ε, Μεσογείου. Να πούμε ποιες είναι οι θέσεις μας. Κάτι το soft όπως λέμε στα γαλλικά, παραδοσιακά. Κάτι το απλό και σας το διαβάζω πολύ γρήγορα. Αρκετά γρήγορα για να το καταλάβουν και οι διερμηνεί. Όχι, αρκετά αργά για να το καταλάβουν οι διερμηνεί. Λοιπόν, σε αυτό το ανακοινοθέν θα λέμε. Η Προεδρία στη συνεδρία τη Βρυξέλλε στο πλαίσιο τη Πολιτική Επιτροπή Ασφάλεια και ανθρώπινων δικαιωμάτων τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Συνοβουλευτικής Συνέλευσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους ή αντέδρασαν ως προς την καθυστέρηση στην εξέβρεση λύσης και ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Συμφωνείτε σε αυτό ελπίζω, δηλαδή όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε. Η κατεπίγουσα ανάγκη για ειρήνη την οποία διεκδικούν ο Παλαιστινιακός και Ισραηλινός λαός οδηγεί τους βουλευτές να ζητούν από τα κράτη-μέλη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τις μεγάλες δυνάμεις αλλά και την Ισραηλινή και Παλαιστινιακή ηγεσία να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανάληψη του διαλόγου. Κοινό αίτημα λοιπόν η επανάληψη του διαλόγου. Και επίσης ζητούν ένταση των προσπαθειών πρωτοβουλειών όπως η τετραμερής στο φύλλο ε, η πρωτοβουλία των Αραβικών κρατών, πρωτοβουλία των ΗΕ και των Ευρωπαϊκών κρατών. Οι εκπρόσωποι των νομοθετικών της νομοθετικής εξουσίας των 32 ευρωπαϊκών κρατών της Ευρώπης και των 11 της ε, ε, Νότιας Μεσογείου καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν, που είναι κοινωνοί της ειρήνης ε, είναι μέλη της ε, Ένωσης για την ε, Μεσόγειο απευθύνουν έκκληση για κάθε δυνατή προσπάθεια που θα οδηγούσε σε ανάληψη του διαλόγου προς την λύση της ειρήνης. Αυτά. Πολύ απλά πράγματα. Απλώς εκφράζουμε τη δέσμευση όλων μας, τη στράτευση των πάντων, στην προσπάθεια για την ειρήνη. Δηλαδή ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις μας να συνεχίσουν τις προσπαθίες τους. Αυτό. Σημειώνουμε ποιες είναι οι τοποθετήσεις μας η Πρόεδρος. Για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα δεν πρόκειται για ψήφισμα αλλά μόνο για δήλωση, για διακήρυξη. Εάν υπάρχουν διαφωνίε, σα προειδοποιώ ότι δεν πρόκειται να περάσουμε μία ώρα να τη συζητούμε. Ο κύριος Σοβιόλζα έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Σα το είπα, εκ των προτέρων σύμφωνα με τα όσα είπε ο συνάδελφος για, για, το ψήφισμα χωρίς να μακρηγορούμε γιατί υπάρχει στο κείμενο πρόβλημα. Δύο προβλήματα. Και είναι θέματα σημαντικά. Πρώτα-πρώτα το ένα είναι θέμα συγκυρία, το άλλο είναι θέμα αρχή. Ότι δηλαδή ένα κείμενο τέτοιου είδου θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από κάποια διακήρυξη, δήλωση, δήλωση κατεβήκοντος χαρακτήρα ούτω ώστε να λέμε ότι όλε οι κυβερνήσεις της ε, Μεσογείου και των θεσμικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, τίθενται αλληλέγγυη με τον Παλαιστινικό λαό, με τον λαό της Γάζας που αυτή τη στιγμή ε, ταλαιπωρείται, βασανίστε πάρα πολύ και δεν είναι δυνατόν να ζητούμε διαπραγματεύσεις, επαφές, ειρηνευτικές κλπ. χωρίς να έχουμε επιδείξει αλληλεγγύη προς εκείνους οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο. Το δεύτερο θέμα είναι περισσότερο θέμα συγκυρίας, διότι είπατε πρόεδρε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα το πρωί. Μα είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν κατάλαβα καλά, ότι ένας αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Πολιτικής της Ευρωμεσογειακή Συνόδου δεν μπόρεσε να έρθει εδώ διότι δεν του έδωσαν θεώρηση στο διαβατήριο. Είναι δυνατόν να ανεχόμεθα κάτι τέτοιο, να μην υψώνουμε τη φωνή μας, ε, προς μια τέτοια κατάσταση. Κάτι το οποίο έπαθε κάποιος συνάδελφος, κάτι το οποίο μας προσβάλλει ως θεσμικό όργανο, ε, ως, ε, ως, σώμα. Επομένως, αυτό θα πρέπει να καταδικαστεί, να καταδικάσουμε αυτήν την αυθαίρετη απόφαση του να παρεμποδιστεί από το να έρθει στις Βρυξέλλες ο συνάδελφος, η πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριο Μπιόλος να διορθώσω, γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Κρέφη έλαβε τη θεώρηση, αλλά του αρνήθηκε η έξοδος από την επικράτεια. Στο ίδιο καταλήγουμε τελικά, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν είναι μαζί μας σήμερα. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ λοιπόν ε, απολύτως μαζί σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σαντούκα. Κύριε Σαντούκα, αλλά σας παρακαλώ σύντομα. Σύντομα γιατί έχουμε ένα ολόκληρο σημείο που μας περιμένει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρόλο που όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές έλαβαν το λόγο χωρίς να τους ζητηθεί να είναι σύντομοι, να πω ότι ο κύριος Δελπίκα συνόψισε την πρωινή μας συζήτηση και όλες τις παρεμβάσεις των συναδέλφων, ιδίω των Ευρωπαίων. Φαίνεται ότι κατάλαβε ότι όλοι επιρρύπτουν ευθύνες στην ε, κυβέρνηση κατοχής του Ισραήλ και τα φρικτά εγκλήματα στην ε, λωρίδα της Γάζας ιδίως. Το ζήτημα λοιπόν είναι σοβαρό. Θα πρέπει όλοι με φωνή ενωμένη να καλέσουμε τους Παλαιστινίους και Ισραηλινούς να εργαστούν στο σκοπό των διαπραγματεύσεων σε συνθήκες ισοτιμίας. Να πω εδώ για την Παλαιστινιακή πλευρά ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που προβάλλουμε φραγμούς. Δεν είμαστε εμείς οι κατέχοντες. Δεν έχουμε εμείς τα κατεύματα κατοχής. Δεν δολοφονήσαμε 1.400 ανθρώπους στην Γάζα, ούτε χρησιμοποιούμε δυνάμεις βίας κατά των Ισραηλινών. Δεν αρνηθήκαμε στους Ισραηλινούς το δικαίωμα να βγαίνουν από τη χώρα τους και να επιστρέφουν σε αυτή. Ο συνάδελφός δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ γιατί τον σταμάτησαν σε σημείο ελέγχου του Ισραήλ. Είναι συνάδελφος κύριε Τελπίκα. Λοιπόν, ξέρω ότι θα το σημειώσετε, αλλά φαίνεται ότι η προσπάθειά σας είναι μια προσπάθεια να αποδυναμώσετε το, τις διαστάσεις του προβλήματος. Εδώ μα ζητάτε στην Επιτροπή αυτή να είμαστε διαφανεί και να αντικατοπτρίζουμε όλε τι συζητήσει που έλαβαν χώρα. Εδώ. Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι λοιπόν κατά τη συζήτησή μας δεν ήταν λιγότερο προσεκτικοί, ούτε λιγότερο ακριβοδίκαιοι. Ήταν σαφή στην τοποθέτησή του. Καταδίκασαν το Ισραήλ και ζήτησαν να πάυσουν οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. Και έφτασαν σε τέτοιο σημείο δεν θέλουμε λοιπόν αποδυνάμωση των διαστάσεων του προβλήματο. Ε, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, λέει ο Πρόεδρο, γιατί οι συνάδελφοι περιμένουν να αρχίσει η συζήτηση για το σημείο 7. Υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να προλάβουν τι πτήσει του. Είναι συζήτηση που έγινε, δεν θα ξαναρχίσουμε. Ο Ρομπέρ θα προτείνει μια λύση, εάν μπορούμε για τη δήλωση. Κοιτάξτε, μια λύση είναι, δεν είσαστε αναγκασμένοι να την εγκρίνετε. Ε, αν μπούμε στι λεπτομέρειε, συμφωνούμε, συμφωνούμε κύριε Σαντούκα. Εάν μπούμε όμω στι λεπτομέρειε, ξαναρχίζουμε τη συζήτηση, δεν θα καταλήξουμε σε καμία απόφαση. Ε, αυτό είναι μια ελάχιστη λύση για να συμφωνήσουμε. Αυτό που μπορώ και προτείνω να προταθεί, έχετε δίκιο για οι δύο, να προσθέσουμε μια τελευταία παράγραφο που να λέει «Η Πολιτική Επιτροπή εκφράζεται τη αρισκιά της για την απουσία του Παλαιστινίου Αντιπροέδρου, ο οποίος δεν έλαβε την ε, ελευθερία να εξέλθει της χώρας». Εντάξει, καταδικάζει αν θέλετε, αντί για τα εκφράζει τη δυσαρέσκειά τη. Θλίβεται και καταδικάζει. Κοιτάξτε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτή θα είναι δήλωση τη Επιτροπή. Ε, ε, αλλιώ δεν θα έχουμε δήλωση. Δεν πρόκειται για ψήφισμα. Δεν, δεν είναι απόφαση για να μπούμε στι λεπτομέρειε έτσι κι αλλιώ. Δυστυχώ δεν θέλαμε να είναι όλα τίποτα, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα έχουμε δήλωση λοιπόν. Πρέπει να σεβαστώ και του συναδέλφου που, που πρέπει να προλάβουν και τα μεταφορικά του μέσα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση, λυπούμε πολύ. Ναι, σταματάμε. Σταματάμε, λέει ο τοπικά. Δεν έχουμε δήλωση, τέρμα. Ναι, είναι περίπλοκο. Τι να κάνουμε, αφού όλοι θέλετε να παρέμβετε τώρα. Όχι, ο στόχος ήταν να εκφράσουμε την άποψή μα, γιατί είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση το πρωί και να αποδείξουμε ότι η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων έλαβε θέση. Είναι απλή δήλωση επί τη αρχή. Το είπε και ο κ. Σομπιόλ. Ελήφθη υπόψη. Ο κ. Σαντούκα ελήφθη υπόψη. Δεν μπορούμε τώρα να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση και να πούμε σε όλε τι λεπτομέρειε θα τελειώσουμε ποτέ. Μια ελάχιστη δήλωση θέλαμε για να μπορέσουμε και εμεί να τη χρησιμοποιήσουμε για τι συνεδρίε του Προεδρείου στι 20 Νοεμβρίου και να λάβουμε θέση και σε σχέση με τα γεγονότα για να καταδικάσουμε την απουσία του Αντιπροέδρου του Παλαιπιστηνίου Αντιπροέδρου που δεν μπόρεσε να λάβει δικαίωμα εξόδου. Κοιτάξτε, ένα λεπτό θα σας δώσω στον καθένα το λόγο. Κύριε Ρέσκι και κύριε Ντάντ, εγώ ήθελα να πειρώσω. Είναι κρίμα να μην έχουμε αυτή τη δήλωση στο τέλος. Ας προσθεθεί το σημείο του για το συνάδελφο που απουσιάζει αλλά νομίζω αυτό που πρέπει να προσθεθεί ούτω ή άλλω είναι το πώ υποφέρει ο λαό τη Γάζα. Μια Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μπορεί να το παραβλέπει αυτό. Νομίζω ότι όλοι θα το δέχονταν αν το λέγαμε κάπου. Αυτό είπε και ο Ραϊμόν. Κύριε Ντάντ, κύριε Αουσδί, ένα λεπτό. Θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου για αυτή την τελική δήλωση, κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε με τρόπο πολιτισμένο το πρωί. Νομίζω οι περισσότερε παρεμβάσει καταδίκαζαν την ε, πλευρά του Ισραήλ. Αυτή είναι η πλευρά που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η, δύναμη κατοχή. Αυτή ακυρώνει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Γιατί να σταματήσουμε και να περιορίσουμε την έκφρασή μα όταν βλέπουμε τέτοια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, αυτή η ισότητα που, για την οποία κάνετε έκκληση με ξαφνιάζει ιδιαίτερω. Πώ να έχουμε προποθέσει ισοτιμία, γιατί να τι έχουμε. Το πρωί καλέσαμε την Ισραηλινή πλευρά να αναλάβει δράση και να αναλάβει τι ευθύνε τη. Και νομίζω ότι και η ευρωπαϊκή πλευρά αυτό πρέπει να κάνει, κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και ποτέ να μην καταλήγουμε σε μια απόφαση. Έφτασε επιτέλου η στιγμή να ζητήσουμε να επιβληθούν κυρώσει. Κυρώσει κατά τη πλευρά που ασκεί βία, που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, που κατέχει τα Παλαιστινιακά και Αραβικά εδάφη. Κυρία Ντάντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πράγματι, η δήλωση αυτή που μας διάβασε ο κύριος Δελπίκα και με όλο το σεβασμό, παρόλο που τον εκτιμώ πολύ, απέχει πάρα πολύ της αλήθειας. Δεν θέτει τα σοβαρότερα ζητήματα, δεν τα εγείρει, δεν τα αγγίζει καν, όπως είπαν οι συνάδελφοι Σαντούκα και ο συνάδελφος από την Ιορδανία. Η δήλωση αυτή μπερδεύει τους ρόλους των του θύματος και του θήτη τους αντιμετωπίζει σαν να ήταν ισότιμοι. Οι απόψει όλων των συναδέλφων νομίζω είναι αντίθετε. Κανεί δεν είπε το πρωί κάτι τέτοιο. Η δήλωση δεν αναφέρει τίποτε. Τίποτε για την κατοχή. Δεν αναφέρει τίποτε για τον Κολάν, για την Ρωσία του Κολάν. Σε μια τέτοια δήλωση, αν θέλουμε να είναι πλήρη, θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η αναφορά. Ιδάλω όχι, α μην υπάρξει. Είμαι κατά. Όχι, όχι, όχι, δεν θα ξαναρχίσουμε τη συζήτηση. Σταματάμε δεν θα έχουμε δήλωση. Συμφωνώ και εγώ. Αλλά σα το είπα από την αρχή. Αν θέλουμε σημεία και λεπτομέρειε, ξαναρχίζει η συζήτηση. Θα καταλήξουμε σε απόφαση ψήφισμα με 30 σημεία. Και δύο ώρε συζήτηση για να καταλήξουμε σε κάτι στο οποίο τελικά κανεί δεν θα διαβάσει. Γιατί θα είναι ένα μακρινάρι. Σταματάμε. Σταματάμε τη συζήτηση. Τα δύο σημεία. Τα δύο σημεία που θα μπορούσαν, αν συμφωνείτε, είναι να διατηρήσουμε το κείμενο. Προσθέτουμε την παράγραφο για την απουσία του Αντιπροέδρου. Καταδικάζουμε και έπειτα μπορούμε να ζητήσουμε το να δοθεί τέρμα στον πόνο και την ταλαιπωρία του λαού της Γάζας. Τώρα, αν θέλετε απόφαση, κείμενο απόφασης με ε, απαρίθμιση σημείων, α, είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ λέω όχι, να μην έχουμε καν δήλωση γιατί ξαναρχίζει η συζήτηση. Δεν γίνεται. Εάν θέλετε λεπτομέρειε θα καταλήξουμε σε απόφαση. Είναι πάντως κρίμα. Κρίμα να μην μπορούμε να, να επιστήσουμε την προσοχή για αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Κοιτάξτε, εγώ θα τη χρησιμοποιούσα για την ε, συνεδρίαση του Προεδρείου και θα την κρατήσω ως δήλωση της Προέδρου Περνάμε στο σημείο 7 λοιπόν τη ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων για την συνεισφορά των εισηγητών. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπω είπα το πρωί, να ευχαριστήσω και του ε, εισηγητέ για την συνεισφορά του. Ποιοτική συνεισφορά. Θα του ζητήσω να παρουσιάσουν τι εισηγήσει του. Έχουμε ένα πρώτο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Ο εισηγητή, ο κύριο Όμπιολ, ο κύριο Χάγκελ ο Ράιντελμαν, ο οποίο ε, ανέλαβε το έργο του προκατόχου, το κύριο Κώστα την Ιταλία δεν παρευρίσκεται σήμερα, δεν θα μπορέσει να παρουσιάσει τη δική του εισφορά. Ο κύριο Ράιντελ λοιπόν και ο κύριο Ρέσγκη. Ο κύριο Ομπιόλσαν ήθελε να ξεκινήσει λοιπόν. Θα είναι πάρα πολύ σύντομη η μου, διότι και η συνεισφορά μου είναι εξίσου σύντομη, εγώ μου ήμουν κάθετα αντίθετο και από ιδεολογική και πολιτική πλευρά προ την ε, η κυρία αυτή, τη Μαργαρίτα, Μαργαρίτα Τσέχ. Και θυμάμαι. Ε, κυρία Θάτσα, συγγνώμη. Ε, θυμάμαι ότι το που μα τα πρώτα δελτία τύπου, εγώ τα πέταγα πάντα στο, στον κάθο των αχρήστων. Πάρα πολύ καλή ιδέα ήταν αυτή και γι' αυτό το λόγο ε, κάθισα και εγώ τώρα και έφτιαξα μόλι, μια μισή σελίδουλα με κάποιε λίγε παραγράφου που μπορώ να το διεξέλθω μέσα σε λίγα λεπτά και δεν χρειάζεται μια ιδιαίτερη εισήγηση. Όμω, αυτό που θέλω να σταθώ έστω και σύντομα είναι ποιο είναι το κίνητρο, ποιο είναι το πολιτικό ελαττήριο τόσο ώστε να φτάσω σε αυτά τα, θέματα τα οποία όμω σα τα είπα προηγουμένω την ώρα που συζητούσαμε τα θέματα τη Ευρωμεσογειακή Ένωση, για να είμαστε λοιπόν ε, ειλικρινεί και ρεαλιστέ. Σοβεί εδώ μια κρίση ε, όσον αφορά την ευρωμεσογειακή πολιτική τη σήμερα ημέρα και θα πρέπει να κάτσουμε και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν θα μπορούσε να πει κανεί μέχρι ότου δεν έχει επιληθεί η, το, το, το, το, Παλαιστινιακό δεν κάνουμε τίποτα. Άλλοι όμως θα μπορούσαν να πούνε ας συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και πάνω στην πορεία θα βάλουμε και εμεί το λιθαράκι μας στην επίλυση της κρίσης. Η δική μου θέση είναι σαφή. Είμαι οπωσδήποτε υπέρ του να συνεχίσουμε την προσπάθεια. πολλέ φορές όταν πάω σε ένα σταθμό του μετρό ή σε ένα πολυκατάστημα και βλέπω ε, μία ε, μία την κυλιόμενη σκάλα μου θυμίζει ακριβώ αυτή την πορεία την Ευρωμεσογειακή. Άμα δεν κάνουμε τίποτα, αν δεν συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε, ε, θα πάμε προ τα πίσω, θα πισωγυρίσουμε. Όπω γίνεται με τη σκάλα αυτή. Επομένω, θα πρέπει να δοθεί στην Ευρωμεσογειακή Ένωση ένα περιεχόμενο πολιτικό μέσω τη πλατφόρμα τη δική μα, τη κοινοβουλευτική. Όμω, από την άλλη μεριά, με ρεαλισμό, α κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε να γίνονται βήματα προ τα εμπρό. Γι' αυτό και εγώ επιμένω σε αυτό το οποίο μου φαίνεται ότι δείχνει σε κάθαρα την κατάσταση. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις στην Μέση Ανατολή. Επομένως, ρεαλισμός είναι ό,τι χρειάζεται περισσότερο αυτή τη στιγμή, διότι αν κανένας έχει κάποιο είδους ε, μαχητικές, ε, ε, ασυμβίβαστες θέσεις, τίποτα δεν θα πετύχει. Θα είναι σαν να μην προχωράει προς τα και επομένως θα έχουμε μόνο πισωγύρισμα. Ε, συγγνώμη αν θεωρείτε ότι σας τα λέω ε, κάπως, ε, κάπως ομά, αλλά αυτό προέρχεται από το ότι ε, νιώθω κάποια κόποση από, από το, το, πώς έγινε η συνεδρίασή μας ε, που δείχνει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Ωραία, αλλά πρώτος και δώσω τον λόγο στον κύριο Ρέντελ, ο οποίος πρέπει να φύγει γιατί πρέπει να προλάβει το αεροπλάνο του. Κύριε Ρέντελ, έχετε λόγο. Äh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θέλω να τοποθετηθώ ως προς το ψήφισμα, αλλά ως προς την έκθεση που πρέπει εγώ να... Όχι τώρα. Όχι για το ψήφισμα. Για το ψήφισμα δεν θέλω να μιλήσω. Για την έκθεση θέλω να μιλήσω. Την έκθεσή μου. Η έκθεσή μου που ζητήθηκε και κατετέθη τον Ιανουάριο του 2009 ε, περιλαμβάνει ένα τμήμα της όλης έκθεσης, δηλαδή αναφέρεται στην προστιθέμενη αξία ε, που προκύπτει για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στην ε, έκθεσή μου που έχετε λάβει εξάλλου στη συνοπτική της μορφή έχω περιοριστεί στα δύο θέματα του ρόλου που μπορεί να διδραματίσει για την περιφερειακή ανάπτυξη όλες τις περιφέρειες εκεί αφενός, αφετέρου δε την κοινοβουλευτική διάσταση για τη ζώνη της Μεσογείου από την ε, Ένωση για τη Μεσόγειο. Για το πρώτο λοιπόν ε, ζήτημα, επιτρέψτε μου γιατί είχα πολύ ε, μεγάλο αριθμό εισφορών ε, προτάσεων για την έκθεσή μου. Να σημειώσω πολύ συνοπτικά ότι είχαμε από την ε, διαδικασία της Βακελώνης σημαντική αναζωγόνηση της κοινωνίας των πολιτών, ενθάρρυνση και ενίσχυση της δημοκρατίας και του ε, δημοκρατικού πλουραλισμού ως στόχο και θα πρέπει και η Ένωση για τη Μεσόγειο να στηριχθεί πάνω στον ίδιο στόχο. Και ως εκ τούτου υποδεικνύω, εάν επιτρέπετε, ότι στην δηλώση των Παρισίων του Ιουλίου του 2008 το γεγονός ότι τα κράτη της Μεσαιουγίου έχουν δεσμευθεί να αναλάβουν να συνεχίσουν τα κεκτημένα της διαδικασία της Βαρκελόνης. Δηλαδή όλα αυτά που συζητούνται σήμερα ήδη έχουν καλυφθεί από την διακήρυξη των Παρισίων. Καθήκον μας ως εκ τούτου θα ήταν εφόσον θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη και αναγκαία η περιφερειακή ανάπτυξη, ως βουλευτές να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ως τμήμα αυτής της ανάπτυξης. το θεωρία όσο και στην πράξη. Για όσα δεν ανέφερε και ο κύριο Κάρλσον και τα σχέδια, τα projects τα οποία, για τα οποία έκανε λόγο, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά απλώ δεν θέλω να πω ότι πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ τη ε, επίσημη, τη τυπική διάσταση που αναλαμβάνουν οι κυβερνητικέ οργανώσει, κυβερνητικοί φορεί, στου οποίου αναφέρθηκε ο κύριο Κάρλσον, και τη δεύτερη διάσταση, ε, το δεύτερο σκέλο, το οποίο εμεί πρέπει να εξασφαλίσουμε, δηλαδή την κοινοβουλευτική ε, διάσταση της διαδικασίας αυτής που παρακολουθεί τα projects αυτά και τα υποστηρίζει. Καθήκον μας είναι κατά την άποψή μου ως εκ τούτου να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και κατά την άποψή μου καλούμεθα ταυτόχρονα μαζί ή παράλληλα με τους ε, επίσημους φορείς ή τους υπηρεσιακούς καλύτερα φορείς να τοποθετηθούμε και ως προς ε, την ύπαρξη ενός ε, φορέα μόνιμης δομής διαρκούς παρουσίας όπως θα ήταν η κοινοβουλευτική συνέλευση αντίστοιχα του ΝΑΤΟ ή άλλων διεθνών οργανισμών με δική της γραμματεία και με δικό της προϋπολογισμό που θα, που χρηματοδοτείται και από τις εισφορές και από πρόσθετα ε, κονδύλια έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα δράσης εμείς ως κοινοβουλευτική συνέλευση, ως βουλευτές. Πράγμα το οποίο συνεπάγεται και πρακτικό έργο και διατύπωση της ε, απέτησης για δικαίωμα ιδίας πρωτοβουλίας σε projects. Επί εταιρικές σχέσεις, ε, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ανοικοδόμηση υποδομών, όλα αυτά τα θέματα τα οποία εξετάστηκαν εδώ, τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά και όχι δεδομένα. Και ιδιαιτέρως σημαντικό και μη δεδομένο είναι το, το καθεστώς του παρατηρητού στις επίσημες ε, εκδηλώσεις τύπου υπουργικές διασκέψεις θα έπρεπε δηλαδή να μας εξασφαλιστεί το, το καθεστώς του παρατηρητή και το δικαίωμα συμμετοχή σε αυτές. Γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική διάσταση στην ε, Ένωση για τη Μεσόγειο. Μεσόγειο. Ωστόσο θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσω την ανταγωνιστική σχέση στην οποία βρισκόμαστε με τον Άτο και τον ΩΣΑ και τους αντίστοιχους φορείς που έχουν αναπτύξει ε, διότι εργαζόμεθα όλοι στον ίδιο χώρο, στα ίδια καθήκοντα και ίσως θα άξιζε τον κόπο να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε περισσότερα σημεία συνεργασίας και επαφής. Δεν ξεκινούμε σε μηδενική βάση, στηριζόμεθα στη διαδικασία της Βαρκελόνης, την οποία εισφέρουμε στην Ένωση για τη Μεσόγειο, την εντάσσουμε στην Ένωση για τη Μεσόγειο και παράλληλα πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση όπως άλλωστε είδαμε και από τις προηγούμενες επικοδομητικές παρεμβάσεις, να παρακολουθήσουμε, να συνοδεύσουμε τη διαδικασία αυτή, διότι έχουμε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο να αναπτύξουμε δράση χωρίς να χρειαστεί να τρέχουμε χωλένοντας πίσω από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Ράιντελ και τώρα το λόγο για ο κύριος Ρεζκή από την Αλγερία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση που μας ζητήθηκε να εκπονήσουμε είχε να κάνει με την εξέταση της προσθέμενης αξίας ε, από την ε, θέση σε λειτουργία, σε ισχύ μάλλον της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Προσπαθώ να κάνω μια σύγκριση στις διακηρύξεις της Βαρκελόνης και των Παρισίων και βέβαια έκτοτε να καταγράψω τα επιτεύγματα. Η διεθνή κοινότητα λοιπόν και κυρίως ε, τα συμβαλόμενα μέρη στην Δέσπης Παρκελώνης ε, σημειώνουν ότι η διαδικασία του 1995 ε, έφτασε στα όρια της σε επίπεδο πολιτικό ιδιαίτερος όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή που δείχθηκε δηλαδή πόσο κρίσιμη και κεντρική σημασία έχει αυτό διότι η κρίση στο Λίβανο αλλά και στη Γάζα ε, οδήγησαν στην, ε, αποτέλεσαν προσκόμματα στην ανάπτυξη της διαδικασία της ε, Βαρκελόνης. Επίσης, τα θέματα της χρηματοδότησης, μάλλον των χρηματοπιστωτικών, αναφέρομαι ιδιαίτερος στο ζήτημα της χρηματοδότησης από το Διεθνές Σημαντικό Ταμείο που δεν αναπτύχθηκε όπως θα περιμέναμε. Και επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διανθρώπινες, διαπροσωπικές επαφές ε, στα κράτη ε, της Βόρειας και της Όχθης Μεσογείου. Το Ίδρυμα αναλύντ και το διαπολιτιστικό διάλογο που όμως δεν μπόρεσε να ε, αποτρέψει την εκτράχυνση των σχέσεων και τις ασυνεννοησίες μεταξύ των πολιτισμών, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε ως παράδειγμα διαβόητη υπόθεση των σκητσογραφιών με τον προφήτη Μωάμεθ που απέδειξαν κατάφορα ότι δεν υπάρχει αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμός τουλάχιστον μεταξύ των περισσότερων κρατών. Επίσης λοιπόν στο πλαίσιο μιας κοινότητας, μιας οργάνωσης, μιας ένωσης κάπως μεσογειακής θα έλεγα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο από το 2005 που ξεκίνησε με την ε, προεδρική παρέμβαση του 2007 από τη Γαλλία και την ε, κήρυξη της Ένωσης για τη Μεσαόγειο στην Ταγκέρη από τον Γάλλο Πρόεδρο το 2007, πλην όμως δυστυχώς ε, δεν ε, έτυχε πλήρους υποστήριξη η πρόταση αυτή, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς αν θέλουμε να προχωρούμε και πρέπει να βρούμε κάποια άλλη λύση και έτσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη δήλωση του Μαρτίου του 2008 ανακήρυξε τη σύσταση μιας ε, ένωσης των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, μιας, ε, και των κρατών της Όχθης Μεσογείου και έτσι ήρθε η ώρα για την Σύνοδο των Παρισίων το 2008. Με τη διακήρυξη των Παρισίων βλέπουμε ε, καταρχά διεύρυνση του αριθμού των μελών από τα 17 ευρωπαϊκά κράτη περάσαμε στα 32 από πλευρά Ευρώπης άρα έχουμε σημαντική εξέλιξη και πάλι βλέπουμε μια ουσιαστική προσθέμενη αξία Η δε αρχηγοί κρατών με τη βούληση να στηριχθούν στο γεκτημένο τη Βαρκελόνη και όχι στην ε, θέση στο ε, στο περιθώριο, ε, επεσήμαναν τη βούλησή του, να αναπτύξουν περισσότερο τι και να μοιραστούν ακόμη περισσότερο τι πολυμερείς ευθύνες. Πέραν των θεσμών ε, που έχει που έχουν προβλεφθεί για την Ένωση, για τη Μεσόγειο, με τη διακήρυξη των Παρισίων προσδιορίζεται η βούληση και συγκεκριμενοποίηση συγκεκριμένων και καθοριστικών πρωτοβουλειών, πάνω από 100 περίπου ε, projects με έξι βασικούς τομείς ε, που αναφέρθηκαν στο προσάρτημα στη διακήρυξη. Και θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα, αν μου επιτρέπετε κυρίες και κύριοι, στους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν συμπροεδρία διετή, έχουμε ετήσια ε, διάσκεψη υπουργών που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα όπως είδαμε διότι η διάσκεψη που είχε προβλεφθεί ανεβλήθη λόγω προβλημάτων στα οποία δεν θέλησε να επιτραφεί ο κύριος Κάρσον. Κοινή γραμματεία ναι, ναι, ναι, ναι. Μα εμείς ξέρουμε γιατί δεν έλαβε χώρα αυτή η διάσκεψη. Και κοινή λοιπόν γραμματεία με εντολή τεχνική η οποία για μας δυστυχώς για μας κατά την διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης 3 και 4 Νοεμβρίου στη Μασαλία αντιμετώπισε δυσκολίες που ε, κάπως ανέφερε ο κ. Κάλσον πολύ περιληπτικά, ένα τα προβλήματα που βλέπουμε εμεί είναι ότι κατακλυζόμεθα από μια σειρά αντιπροέδρων και αναπληρωτών γραμματέων. Και βέβαια ένα ζήτημα που δεν έχει επιληθεί ακόμη είναι το καθεστώ. Η σύσταση λοιπόν ήταν να υπάρξει ένα καθεστώ, το οποίο θα ε, ορίζεται με βάση κριτήρια αποτελεσματικότητα και νομιμότητα νομιμοποίηση και έτσι το ότι έχουμε τόσους πολλούς ε, φόκους, τόσες πολλές θέσεις αναπληρωτών γραμματέων μας οδηγεί στην ανησυχία, μας γράφει την ανησυχία ότι θα παρασυρθούμε προς ένα πολιτικό όργανο περισσότερο παρά ε, προς την έννοια της ε, Γενικής Γραμματείας. Αυτά. Θα μιλήσω περισσότερο από ότι ο κύριος Ράιντελ για την κοινοβουλευτική συνέλευση ε, επίσης ακούστηκαν κάποιες άλλες παρατηρήσεις ως προς την κοινοβουλευτική συνέλευση, η οποία τίνει να μετατραπεί σε κοινοβουλευτική συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο παρά το παρελθόν της και αφήνω στην άκρη της, ε, της συνάντησης στη Βαλενσία, της Νάπολης, την διάσκεψη, όλα αυτά τα οποία επισήμαναν και οι προκάτοχοί μου και που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια και υπενθυμίζω την διακήρυξη της νεκράς θάλασσας που ζητήσαμε να, καθιστού, να καταστεί η, η κοινοβουλευτική συνέλευση το κοινοβουλευτικό στέλος, σκέλος της Ένωσης για την Ευρώπη, για τη Μεσόγειο, συγγνώμη, που όμως παρά τις διακηρύξεις αυτές και όλο το παρελθόν και όλη την ιστορία, την πορεία που έχουμε χαράξει, απεφάσισαν οι υπουργοί στη Μασαλία τελικά να αγνοήσουν τις ε, προτάσεις μας και να ε, δηλώσουν μόνο ότι χρειάζεται να βελτιωθούν οι σχέσεις της κοινοβουλευτικής συνέλευσης με τους εταίρους της μέσα σε όλη τη διαδικασία. Άρα λοιπόν αντί να καθιστούμε αντί να καταστούμε μια πραγματική κοινοβουλευτική συνέλευση και να μπορέσουμε να ε, συμβάλλουμε στην ε, Ένωση για τη Μεσόγειο και την επιτυχία της με βάση τα, ε, των Παρισίων περιοριζόμαστε σε μια συνοδευτική μόνο θέση, ένα συνοδευτικό μόνο ρόλο. Επίσης σήμερα ότι υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι θα έλεγα όχι απαραίτητα ότι είναι ανταγωνιστικοί, αλλά πάντως έχουμε επικάλυψη αρμοδιοτήτων και έργων και μια είναι εδώ και η ε, φίλοι από τη Μάλτα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην στην ύπαρξη της ΠΕΜ ε, και όχι μόνο της ΑΠΕΜ. Έτσι λοιπόν έχουμε όργανα τα οποία αντικαθιστούν το ένα το άλλο ε, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τα λοιπά κοινοβούλια έχουμε εκπροσώπους και στα δύο όργανα και αυτό σημαίνει λίγο πολύ ότι κάνουμε την ίδια δουλειά. Όταν ε, μέσα από μία στιγμή ενδεχομένω απόφαση αποφασίσουμε την ε, Ευρω... τη Μεσογειακή Διάσκεψη να τη μετατρέψουμε σε Ένωση για τη Μεσόγειο και την Ένωση για τη Μεσόγειο να την μετατρέψουμε σε Ευρωμεσογειακή Ένωση, τα πράγματα περιπλέκονται πολύ και ιδιαίτερα για τα ανθρωπιστικά. Όλα τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, είναι περίπλοκα, υπάρχουν ζητήματα χρηματοπιστωτικά και οικονομικά πολύ δύσκολα. Βέβαια πάνω από όλα έχουμε το ζήτημα τη ε, σύγκρουση στο το μεσανατολικό δηλαδή που έχει γνωρίσει δύο τεράστιες κρίσεις έχει οδηγήσει στην ε, βραδιπορία προς τη θέσπιση των ε, δομών και την καθυστέρηση σε όλα τα σχέδια γιατί εφόσον δεν υπάρχει και γραμματεία ε, δεν μπορούν να αναπτυχθούν τα σχέδια. Γνωρίζουμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα ύστερα από την τελευταία στιγμή, την τελευταία στιγμή ματέωση των, ε, της συναντήσεως των ΕΠΑ των, ε, των αξιωματούχων το Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες, τα προβλήματα σχέση με τον Αραβικό Σύνδεσμο, διαφορές που οριστικά πλέον διευθέτησαν οι Υπουργοί μετά είχαμε μια τελευταία κρίση τώρα το, Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο του τελευταίου, ύστερα από τις επιθέσεις βάρος της Λορδίας της Γάζας όπου σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. Και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί μια ρύθμιση οριστική, δίκαιη, βιώσιμη, ε, της ε, σύγκρουσης μέσα από τις διάφορες ε, διαδικασίες, τις πρωτοβουλίες των αραβικών κρατών, την αντιμετώπιση των προκλήσεων σταθερότητας και ασφάλειας που αντιμετωπίζει κυρίως η Ανατολική Μεσόγειος, χωρίς την οποία, υπογραμμίζω χωρίς την οποία, η οδήποτε πρόοδος ως προς την ανοικοδόμηση και την εταιρική σχέση, ως προς την ασφάλεια και την σταθερότητα δεν μπορεί να νοηθεί. Η αντιμετώπιση της αραβικής σύραξης δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητα από την Ένωση για τη Μεσόγειο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να λυθεί η ε, Ισραηλινο-Αραβική διένεξη για να δημιουργηθεί η Ένωση για τη Μεσόγειο. Όχι, τα πάντα πρέπει να επιδιώξουμε να τα επιτύχουμε ταυτόχρονα. Τα προβλήματα και εμείς εδώ ως βουλευτές ε, τα γνωρίζουμε τα βλέπουμε καθημερινά στη τελευταία ανάλυση για να έρθουμε σε ένα ταξίδι εδώ στην Ευρώπη. Καθημερινές δυσκολίες έχουμε, περνάμε από χιλιάδες ελέγχους και σε τούτου η περιστολή των, της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των ε, οχθεών της Ευρώπης είναι ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, να απελευθερωθεί η κίνηση πολιτών μεταξύ των δύο όχθεων έτσι ώστε να σταματήσουν αυτές οι κατασταλτικές πολιτικές, να γυρίσουμε πίσω στη διάσκεψη των Παρισίων, να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών για να προσεγγίσουμε ένα τον άλλον και να καταλάβουμε ένα τον άλλον καλύτερα. Το Ίδρυμα Αναλίντ φυσικά είναι ε, είναι ίδρυμα Euromed, Euromed, όχι μεταξύ δηλαδή Σουηδίας και Αιγυπτού, αυτό το γνωρίζουμε όλοι, δεν υπάρχει λόγο να το επαναλαμβάνω. Ε, τα δε σχέδια αν επιτρέπετε για να κλείνω, χρειάζονται συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Η διαδικασία επιλογή των επιλέξιμων σχεδίων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στου όρου τη ειρήνη, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να λαμβάνει υπόψη τον περιφερειακό, υποπεριφερειακό και δια ε, συνοριακό ή διεθνικό χαρακτήρα καθώς και την διασυνδεσιμότητα των διαφορών περιφερειών. Η μεταβλητή γεωγραφία όπως ε, προτείνει η Αλγερία θα επιτρέψει σε κράτη-μέλη που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ τους ή είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους να βοηθήσουν και να υποβοηθήσουν τη διαδικασία αυτή. Προβλήματα όπως η ρήπαση της Μεσογείου, ε, το ηλιακό σύστημα για τη Μεσόγειο οι αυτοκινητόδρομοι της ε, θαλάσσης μπορούν ε, να αποτελέσουν ε, φάρους στην διαδικασία αυτή με επιλογές αντικειμενικές που όμως δυστυχώς ορισμένα κράτη-μέλη προτίμησαν να θέσουν στο περιθώριο με την συνωμοτική στάση κάποιων άλλων πρέπει να πω που οδήγησαν σε καθυστέρηση και αποτυχία κάποια από τα σχέδια. Η έλλειψη συντονισμού από πλευράς Ευρωπαϊκής η οποία, ο συντονισμού οδήγησε και σε προβλήματα στην διάσκεψη των Παρισίων και την απουσία συμμετοχή των αραβικών κρατών. Πρέπει επίση να σημειώσουμε ότι η οικονομική διάσταση στη ζώνη έχει πολύ περιορισμένε δυνατότητε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μόνο 2% των επενδύσεων τη στα κράτη τη Νότια Όχθη Μεσογείου, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν περίπου 20% των επενδύσεων ή και περισσότερο. Ε, οπότε άλλωστε είπε κάποιο από του συμμετέχοντε τη των Περισσίων και το ακούσαμε και σήμερα το πρωί από κάποιον ομιλητή, η Ευρώπη στηρίχθηκε στην ΕΚΑΧ, η Ένωση για την Μεσόγειο θα πρέπει να στηριχθεί στον ήλιο και τη θάλασσα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσθέμενη αξία από την Ένωση για τη Μεσόγειο που θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, μια πρωτοβουλία σημαντική με ανάγκη για σταθερή υποστήριξη. Η δική μου χώρα η οποία έχει πρώτο στατήσει στην ε, σύσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο με την αποφασιστική της συμμετοχή και την υποστήριξη από πλευρά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Διασκέψεως των Παρισίων πιστεύει ότι ανεξαρτήτως της μορφής που θα λάβει αυτή η νέα εταιρική σχέση μεσογειακή ή ευρωμεσογειακή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια ένωση στέρεη μια ένωση βιώσιμη με εταιρική σχέση μεταξύ τη ε, βόρεια και τη νότια όχθη Μεσογείου, όπου όμω η νότια όχθη θα έχει τη θέση που τη αξίζει και που θα μπορέσουμε έτσι να οδηγηθούμε σε μια μηδέα κατανόηση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ρασκή. Την παρουσίαση αυτή για όλα αυτά τα ζητήματα τη θεωρούμε πολύτιμη. Κύριε Βάγγελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να πω δύο λόγια και ελπίζω ότι θα παραμείνω ακριβώς σε δύο λόγια. Η σημερινή συνάντηση θυμίζει τη Μεσόγειο θάλασσα μετά από τρικυμία, μετά από μια μέρα καταιγίδα. Έχουμε λίγα παγόβουνα από τη Σουηδική Προεδρία και τους Γερμανούς συναδέλφους αλλά μπορούμε να συζητήσουμε και με ηρεμία και φιλήσυχα. Θα πρέπει ως νέος μέλος του Κοινοβουλίου να πω ότι με συναρπάζει η σημερινή συζήτηση η οποία δείχνει τι καλές ευκαιρίες έχουμε αλλά και τι ευθύνες προκειμένου να φέρουμε το διάλογο και να έχουμε επικοδομητική συζήτηση στην ε, Μεσόγειο για τους σκοπούς της ευρωμεσογειακής σχέσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον ε, κύριο Κάζεκ όπως αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε διότι παρέλαβα το έργο του. Είμαι ο κληρονόμος του και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που μπορώ τα περισσότερα από τα ευρήματά του και τα πορίσματά του να τα συμπεριλάβω στην δική μου τη συνεισφορά. Να τονίσω ότι η σημερινή συζήτηση για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και η πρόσφατη συζήτηση για την έκθεσή μας δείχνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας αναζητώντας μια θετική επίλυση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής ένεξης. Δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες για το κατά πόσον δεν θα πρέπει να είμαστε δέσμοι του προβλήματος, ίσως και να μην επέλεξα για τους σωστούς όρους. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι σαφώς σοβαρότατο, όμως θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να διευρύνουμε, να εμβαθύνουμε το διάλογο με συγκεκριμένα προγράμματα, προγράμματα που να υλοποιηθούν στην περιοχή της Μεσογείου. Και να μην απαρνηθούμε, να μην παραβλέψουμε τις βασικές αρχές του δικαιώματος του κάθε ανθρώπου, του κάθε έθνους στην ελευθερία, στην ελευθερία της έκφρασης, στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα να χτίσει το δικό του ελεύθερο κράτος, ανεξάρτητο κράτος, μιλώντας για τους Παλαιστινίους. Επίσης, ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την Ένωση για τη Μεσόγειο ως ευκαιρία, ως πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε διάλογο στα πλαίσια μιας νέας δομής και να φέρουμε κοντά 44 χώρες που συμπεριλαμβάνουν όλους τους εταίρους που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν στην ίδια αίθουσα, γύρω από το ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Να δημιουργήσουμε επίση έναν μηχανισμό για τη διαχείριση κρίσεων αξιοποιώντας και την Ένωση για τη Μεσόγειο και εντατικοποιώντας τις σχέσεις για την μέτρηση των διενέξεων και την επίλυση των σειράξεων. Να ευχαριστήσω όσους τόνισαν ότι κατεπήγει η ανάγκη της δημιουργίας της Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο, ώστε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα να υπερπηδήσουμε τις δυσκολίες με συγκεκριμένα και χειροπιαστά προγράμματα διμερούς και πολυμερούς συνεργασία. Άλλο ένα πόρισμα που αφορά την Ένωση Μεσόγειο είναι το εξή, ότι η ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Οπότε θα ενισχυθεί η δημοκρατική της ε, νομιμότητα για να, για να γίνει αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα δομή της κοινοβουλευτικής ευρωμεσογειακής συνέλευσης. Θα πρέπει να είναι προσκεκλημένη τουλάχιστον ως παρατηρητρία και να εκφράζει τις κυβερνήσεις ε, και επίσης να προετοιμάζει τις συναντήσεις των ε, ανώτατων εκπροσώπων. Να θυμίσω επίσης ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο συμπληρώνει και δεν είναι εναλλακτική διαδικασία για την ε, σχέση της ε, ένταξης για τις χώρες που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία και έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κλείσω εδώ. Διαβάστε την έκθεση και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Σαντούκα. Και θα πρέπει να κλείσουμε κάποτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι όσο τηλεγραφικός γίνεται. Όμως θα χάσω μια εβδομάδα τον ύπνο μου αν δεν μπορούσα να σας πω τι πιστεύω όσον αφορά αυτά που ελέγχθησαν. Εγώ πάρα πολύ συγχυστή όσον αφορά κάποιε απόπειρε ορισμένων να, να περάσουν έτσι επιδερμικά το πρόβλημά μα να ψεφτάξουν ένα ξεροκόμματο ε, και έτσι να τα κουκουλώσουν. Ο Χασάν Χρήσα είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα ε, στέρηση ελευθερίας. Πρόκειται για ένα μικρό κομματάκι του μεγάλου μεγάλου προβλήματος. Παρακαλώ να μην θεωρείτε ότι αυτό είναι μικρό πρόβλημα, να το δείτε στους πραγματικούς euh, Πρόεδρος. Για τον κύριο Κρέισι θα κάνω εγώ μια δήλωση. Θα προβώ εγώ σε, κάποια, σε σύνταξη επιστολής που θα διαβιβάσω αρμοδίως στις Παλαιστινικές Αρχές τόσο ώστε να τους πω ότι καταδικάζουμε το ότι ένας αντιπρόεδρος μας δεν μπόρεσε να έρθει να συμμετάσχει στις εργασίες της Επιτροπής μας. Θα πάει αυτό και στις Ισραηλινές αρχές για τον ε, κύριο αυτό που είναι μέλος του Προεδρείου της Ευρωμεσογικής Διάσκεψης. Και τώρα, πάμε στο δεύτερο θέμα. Ευχαριστώ τους ε, εισηγητές όσον αφορά την ε, Ένωση. Το δεύτερο θέμα ήταν η ελευθερία έκφρασης όσον αφορά τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως είπε η κυρία Φλότρο. Ε, κυρία, μια κυρία συνάδελφος τέλος πάντων, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι είπε ο καθένας, ναι. αλλά και το έργο το οποίο επετέλεσαν από κοινού. Θα δώσω όμως την κυρία Φλότερο τώρα το λόγο, τόσο ώστε να μας πει τι έχει για το θέμα εκείνο. Έχουμε, όπως μας είπατε κυρία Πρόεδρε, αυτή μας την προσπάθεια του να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική θέση που αφορά ε, αυτό το σχέδιο το οποίο ε, θα πρέπει να συζητηθεί και έχουμε κάποιες γενικές αρχές και πάρα πολλοί θεμελιώδεις που είναι οι εξή. Όπως μπορείτε στις τις παραγράφους ε, από α έως ζ επενθυμίζουμε ποια είναι τα μέσα του διεθνούς δικαίου τα οποία ρυθμίζουν τα της ε, ελευθερίας έκφρασης και τα του δικαιώματος στην ε, ελεύθερη και θρησκευτική πίστη στη συνέχεια. Όπως ξέρετε, πολλές φορές σε κάποια δημόσια συζήτηση ε, υπάρχουν κάποια όρια, ας πούμε, το ότι θα πρέπει να πούμε ότι η ελευθερία της θρησκείας είναι και η ελευθερία, το δικαίωμα στην αθεία ούτως πίστη στο να μην έχει κανείς σκεφτική πίστη ή και στο δικαίωμα του να μπορεί να αλλάξει κανείς θρησκεία. Κάτι άλλο για αυτό το συμβαστικό κείμενο, το οποίο υπάρχει προσζήτηση είναι ότι αυτές οι δύο ελευθερίες είναι δυνατόν να συζητηθούν και να γίνουν αντικείμενο Εκμετάλλευση από κάποια μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, να <clears throat> είναι αντιφατικές αυτές οι δύο ελευθερίες σκέψη ή σκεφτικής πίστης γιατί σε, κάποια, ε, σε κάποιες καταστάσεις, σε σε κάποια κράτη που έχουμε κάποιο θρησκευτικό φανατισμό, το ότι αυτό φημώνει την ελευθερία τη σκέψη. Από υπάρχει και αυτή η αντίληψη περί του ανταγωνισμού, του αντίφαση αυτών των δύο δικαιωμάτων. Εμεί όμως θέλουμε να πούμε πόσο είναι ελεύθερα μεταξύ τους. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Είναι αλληλεξαρτώμενα. Στην πραγματικότητα η άσκηση του ενός δικαιώματος ενδυναμώνει το άλλο. ένας ενάρετος κύκλος της αμοιβαίας ενίσχυσης των δικαιωμάτων αυτών. Έκφραση, σκέψεις, σκέψεις θρησκευτικής ελευθερίας. Βεβαίως, δεν πρέπει κανείς να είναι αφελής, θα πρέπει κανείς να τονίσει ότι αυτά τα δικαιώματα δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα, δεν έχουν όρια, δεν ασκούνται εν κενό, θα πρέπει να ασκούνται με υπευθυνότητα. Ακριβώ όπω προβλέπει το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων, την των Δικαιωμάτων. Υπάρχει ολόκληρη νομολογία όσον αφορά την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης. Ότι όταν η ελευθερία της έκφραση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη, τότε προβλέπει η Επιτροπή των Δικαιωμάτων ότι υπάρχουν κάποιε θεμητέ, ε, θεμητοί περιορισμοί που πρέπει να τεθούν. Άρα δεν πρέπει κανείς όλα αυτά να τα αντιλαμβάνεται με συναισθηματική φόρτιση. Ή να επηρεάζεται από κομματική τοποθέτηση. Θα πρέπει κανεί να τα βλέπει αυτά αμερόληπτα. Όπω γίνεται από κάποιο όργανο τη δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα να πούμε και συμπληρωματικά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το πόσο σημαντικό είναι το να ασκείται ως πολιτική καταπολέμηση του ρατσισμού. Γιατί μόνο με την ανεκτικότητα είναι δυνατόν να προστατεύσουν αυτά τα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την ευρωμεσογειακή υπόθεση. Πολλές φορές υπάρχει παρεξήγηση, παρανόηση. Πολλές φορές γίνεται συζήτηση αυτών των θεμάτων με συναισθηματική φόρτιση. Αυτά όσον αφορά τα δικαιώματα, όσον αφορά την ομολογία. Και όσον αφορά την κατανόηση, θα πρέπει να γίνει όσον αφορά το πώ ασκούν αυτά τα δικαιώματα ε, στον ιδιωτικό χώρο και στο δημόσιο βίο. Βεβαίως και όλα αυτά επιδέχονται βελτίωση, επιδέχονται εμπλουτισμό. Βεβαίως και οι συνεισηγητές μείναμε σε αυτές τις δύο σελίδες που είπε και ο κύριος Σομπιόλς. Οπότε να τα συζητήσουμε, να προβληματιστούμε με αφετηρία αυτές μας τις προτάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Ντάκη τώρα. το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι. Σήμερα, σε σχέση με αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, εμείς μπορούσαμε μόνο να δουλέψουμε πολύ σύντομα. Θα ήθελα απλώς, όσα είπαν ε, στα όσα παρουσιάσαμε την έκθεσή μα, να παρακαλέσω του ε, κυρίε και κυρίου συναδέλφου αν έχουν κάποια παρατήρηση, κάποια συμπλήρωση. Πολύ ευχαριστώ να την ακούσουμε. Ω προ την ελευθερία τη έκφραση, ω προ την ελευθερία τη θρησκευτική πίστη, βεβαίω ε, ακόμη και αν κανεί βλέπει τα πράγματα αυτά με διαφορετικό μάτι, ξέρουμε ότι μετά τον, ε, το πέρα του ψυχρού πολέμου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ουσιαστικό πρόβλημα Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν δομέ οι οποίε δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτέ τι δυσκολίε, διαρκώ μεταβάλλονται και μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου για λόγου ψυχολογικού και άλλου. Ε, αντιμετωπίσαμε συγκρούσεις οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκληθεί από τις ρήξεις του ψυχρού πολέμου. Ένα παράδειγμα ήταν ε, η, η κρίση με τις γελιογραφίες εις βάρους του ε, προφήτη Μωάμεθ. Αυτό ήταν ένα πολύ σαφές ε, παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διαφοροποιούμε, ως προς τη θεώρηση της ελευθερίας. Διότι ελευθερία δεν μπορεί να είναι μεμονωμένη ελευθερία. Έχουμε να κάνουμε με ένα όλο ένα σύνολο ελευθεριών. Δεν μπορούμε να βάζουμε χωριστά στο κάνσολο την κάθε ελευθερία και να λέμε πότε πότε είναι θεμελιωμένο το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και πότε πότε δεν είναι γιατί τότε μόνο προβλήματα μπορούμε να έχουμε. Ιδιαίτερα δε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μετά την κρίση στο Ιράκ, μετά την κρίση στο Αφγανιστάν, μετά την ε, συνεχιζόμενη όλα αυτά τα χρόνια ε, διαφορά, σύγκρουση μεταξύ Ισραηλών και Παλαιστινίων βλέπουμε ότι πρέπει να διερευνήσουμε νέους δρόμους για την αναγνώριση των ελευθεριών ε, των μεν και των δε. Με πολύ μεγάλη προσοχή και, και φρόνηση. διότι βλέπουμε ότι οι κοινωνίες μας είναι ευάλωτες, μπορούν να πάσα στιγμή να κινητοποιηθούν και να, ε, να οξυνθούν τα πνεύματα, να βρεθούν αντιμέτωπες η μία απέναντι στην άλλη και ε, να αντιμετωπιστούμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Το βασικό λοιπόν δεν είναι ποιο έχει την πλειοψηφία, ποιο ε, μπορεί να επιβάλλει τη γνώμη του στον άλλον, αλλά το ε, πώ θα εξασφαλίσουμε τον πλουραλισμό, το σεβασμό δηλαδή των πάντων. Η ελευθερία της θρησκευτική πίστης είναι αλληλένδετη ρηκτά με την ελευθερία της έκφρασης αυτό σημαίνει και σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης αλλά και σεβασμό στη σκεφτική πίστη, δηλαδή αποτροπή ε, περιστατικών και κρίσεων όπως αυτή των γελιογραφιών εις βάρος του προφήτη Μωάμεθ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο θα λάβει ο κύριος Πεντρέτς. Όσο πιο σύντομα θα πω πρώτα. Πρώτα πρώτα, συμφωνώ 100% με τις παρεμβάσεις των δύο συναδέλφων που έλαβαν τον λόγο. είχαμε φετηρία τρία έγγραφα. Τελικά ήταν σύμβατα μεταξύ τους. Και καταλήξαμε σε σύνθεση. Όσον αφορά αυτόν τον συμβιβασμό σε ένα κείμενο το οποίο και σας υποβάλλουμε. Διαπιστώθηκε ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης και όσον αφορά ε, τις σχετικές πίστης και από την άλλη μεριά φρία της έκφρασης ε, είναι συμβατά δεν αντιμάχεται το ένα το άλλο δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει αιτία να συγκρούνται μεταξύ τους αυτά τα δικαιώματα προτείνουμε το πώς έρονται οι σχετικές αντιφάσεις και συγκρούσεις και είπαμε σε τι επίπεδα θεωρήσαμε τα διάφορα θέματα, ούτως ώστε να καταλήψουμε αυτές τις προτάσεις και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ανοχή, εκπαίδευση, ε, ενημέρωση του ενός για την κουλτούρα του άλλου και δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να υπάρχει κάποιο είδος περιορισμός της έκφρασης πέραν των ορίων που πηγάζουν από την άσκηση των υπολείπων δικαιωμάτων. Είπαμε επίσης το ότι θα πρέπει όχι με καταστολή αλλά με εκπαιδευτικό τρόπο κανείς να διαδίδει να υποστηρίζει αυτά τα δικαιώματα. Και βεβαίως όπως πάντα δουλεύουμε στην Ευρωμουσιακή Ένωση θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ούτως ώστε να επιφέρουμε ότι βελτιώσεις ε, προταθούν και να προχωρήσουμε έτσι στο μέλλον. Θέλετε κύριε Σαντούκα κάτι να πείτε πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις θρησκείες, έχω να σας πω τα εξή. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Γιατί όλες οι θρησκείες πρεσβεύουν κάποιες αξίες υψηλές, ελευθερία, ανεκτικότητα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τις θρησκείες. Το πρόβλημα αναδύεται όταν κάποιοι θέλουν να τις εκμεταλλευτούν πολιτικά τις θρησκείες, θέλουν να τις έχουν ως όχημα, ούτως ώστε να καταφέρουν κάτι σε κάποιο επίπεδο, ατομικό, τοπικό, να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα. Δηλαδή. Εμείς έχουμε υποφέρει ακριβώς από τέτοιου είδους ε, ε, χρησιμοποίηση της θρησκείας. Και έτσι καταλήξαμε να παλεύουμε να χάσουμε, να, να δικινδυνεύουμε, να χάσουμε τη γη των προγόνων μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα στην κυρία Φλότρο για τόσα ανέπτυξη όσον αφορά την ελευθερία της ε, έκφρασης και σε σχέση με τα όσα είπε για τα όρια της ελευθερίας ε, που είναι η άσκηση των υπολείπων δικαιωμάτων. Έχουμε και εκείνα τα σκίτσα βεβαίω. Τα σκίτσα αυτά κυκλοφόρησαν με αφορμή, με πρόφαση την ελευθερία της έκφρασης. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος Ευρωπαίος ιστορικός γράφει για το ολοκαύτωμα και κάτσει και πει ότι Φερρυπίν το ολοκαύτωμα ε, υπήρξε ή δεν υπήρξε. Όμως από την άλλη μεριά φουσκώνουν τον αριθμό των ε, θυμάτων. Τι γίνεται τότε με αυτό τον ιστορικό. Σύρεται σε δικαστήρια στην Ευρώπη. Αν γίνεται κάτι τέτοιο, τότε δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση που να μπορεί να ασκήσει αυτός ο συγγραφέας. Όταν όμως αυτό αφορά άλλου λαούς, τότε λέμε ναι υπάρχει αυτή έκφραση. Υπάρχει δικαίωμα ο καθένα να εκφραστεί γνώμη του. Άρα εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και εδώ είναι το πρόβλημα. Εμεί που ότι διάσταση των δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να προσβάλλει κανέναν. Εμεί ερχόμαστε από τη Μέση ε, υπάρχουν πολλοί θρήσκοι και όπως υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι θρήσκοι πρεσβεύουν κοσμική αντιμετώπιση. Περισσότεροι είναι θρήσκοι πάντως που θα συμφωνούσαν. Ότι δεν θα πρέπει κάτι να υποθεί ούτως ώστε να προσβάλλει είτε τον Χριστό είτε τον ε, Μωάμεθ ή την Παναγία. Γιατί πιστεύουν ότι και ο Χριστός αλλά και ο Μωάμεθ από τη δική μας περιοχή του κόσμου προέρχονται. Πιστεύουν σε, σε, ε, σε αυτές τις ε, αξίες. Γιατί πρόκειται για πολιτισμό, πρόκειται για κουλτούρα, πρόκειται για αξίες με τις οποίες ζήσαμε πολλούς αιώνες. Ακόμα και οι άθεοι, ακόμα και οι μη θρήσκοι. Και θεωρούμε ότι και ο μαμαθικείο Ιησούς συνέβαλαν στην πρόοδο της ανθρωπότητας. συνέβαλαν στην, στην κατοχήρωση κάποιων αξιών. Επομένως, αυτό θα πρέπει να το σπαστούν όλοι, όχι μόνο ένας μουσουλμάνος η ένας χριστιανός. Δεν πρέπει να, να προσβάλλεται η Παναγία ή ο Ιησούς ή ο Μάμεθ. Άρα θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, να γίνει αντιληπτή με θετικό τρόπο η ελευθερία της έκφρασης. Και όχι με αρνητικό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που δυνάμει μπορεί να προσληφθούν και πολλές θρησκείες. Ευχαριστώ κύριε Σαντούκα. Άλλες παρεμβάσεις. Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι η ελευθερία της έκφρασης ταυτίζεται απολύτως με την έννοια της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να διαχωριστεί από αυτήν. Ένα ανθρώπινο είναι το ίδιο είτε βρίσκεται στο βορρά είτε στο νότο είτε στην Ασία είτε στην Αφρική. Είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα. Πώς λοιπόν να εξηγήσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα σεβαστούμε όταν βλέπουμε να παραβιάζονται συνεχώς. Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία έκφρασης από δυνάμεις κατοχής, κατακτητικές δυνάμεις κατοχής. μετά από όλες αυτές τις πράξεις κατά των ανθρώπων αυτής της χώρας, πώς μπορούμε να μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τιμωρώνται μπροστά μας οι Παλαιστίνοι, όταν σήμερα δεν έχουμε δικαίωμα να προβούμε σε ελεύθερε δηλώσει για το τι του συνέβη. Πού είναι η ελευθερία τη έκφραση, Δεν είναι ντροπή. Ντροπή να φύγουμε από αυτή τη συνεδρίαση χωρί τη δήλωση που προηγουμένω ακούσαμε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να έχουμε μια τέτοια δήλωση όπως αυτή που ετοίμασε όμως η γραμματεία και τελικά καλύτερα να μην ε, προκύψει κάτι τέτοιο από αυτή τη συνάντηση. Αυτό που κάνει το Ισραήλ στα Παλαιστινιακά δάφη ονομάζεται φρικαλαιότητα. Είναι πράξεις βίας κατά των ανθρώπων αυτή τη χώρα και θα συμφωνήσω με την, Τουρ... με Τουρκάλα αυτό που είπε. όλα τα συντάγματα όλων των κρατών της Φιλίου και οι δηλώσεις του ΟΗΕ εξασφαλίζουν την ελευθερία της έκφρασης και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά άσχετα από το φίλο, την εθνικότητα ή το, τη θρησκεία. Πώς όμως να εξηγήσουμε ότι 5 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αυτής υποβάλλονται σε κάθε είδους διακριτική μεταχείριση. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Σαντούκα, είπε στις χώρες μας με μονοθεϊστικές θρησκείες, στο χριστιανισμό, μάλλον ο χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός και ο μεθανισμός προήλθαν από αυτή την περιοχή. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, δυνατο... δεν... δυνατότητα να αποδεχτούμε την διακριτική μεταχείριση λόγω θρησκευτικών επιθύσεων. Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο που στο Σύνταγμά τους ήδη προβλέπουν επιλέξει ότι απαγορεύεται να προσβάλλεται ο επικεφαλής της χώρας, η βασίλισσα λόγου χάρη ή οποιοδήποτε κατέχει την εξουσία λόγω της ελευθερίας της έκφρασης. Αλλά κάποιες χώρες προβλέπουν το συνταγμά του την απαγόρευση προσβολή του ολοκαυτώματο λόγου χάρη. Υπάρχουν ιστορικοί, υπάρχουν επιστήμονε που μελέτησαν το θέμα αυτό και δικάστηκαν όταν διαφώνησαν με τι γενικέ τάσει και απόψει. Δεν θα έπρεπε οι χώρε αυτέ που προβλέπουν κάτι τέτοιο στο Σύνταγμά του να θεσπίσουν και νόμου. Νόμου που να προσάγουν σε δίκη όσους προσέβαλαν άλλους ε, με την δικαιολογία της χρήσης της ελευθερίας της έκφρασης, της άσκησης μάλλον της ελευθερίας της έκφρασης. Διότι η ελευθερία της έκφρασης μπορεί να μας δημιουργήσει στο χάος, ένα δημιουργικό χάος το χρησιμοποίησε και η κυβέρνηση του κυρίου Μπούς. Όταν λοιπόν η ελευθερία της έκφρασης δεν δημιουργεί συγκρούσεις μεταξύ των λαών, ναι, να χρησιμοποιηθεί και να ασκείται, αλλά όχι να είναι δικαιολογία για εξτρεμιστές να συνεχίζουν τις δράσεις τους, τις επέσχετες δράσεις τους, να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό και να σεβόμαστε τις θρησκευτικέ οπιθήσεις του καθενός, να τη βλέπουμε τις θρησκείες στο σωστό του πλαίσιο. Ε, θα ζητήσω από τους συναδέλφους που ασχολούνται με την σύνταξη των νόμων, θετικών κειμένων και την έγκρισή τους, να φροντίσουν σε αυτά, να διασφαλίζουν και τους ανθρώπους και το σεβασμό των χωρών, άσχετα με τις θρησκευτικές οπιθήσεις ώστε να αποφύγουμε όλους τους αρνητικές συνέπειες από τέτοιες δράσεις. Ευχαριστώ κύριο Δερπικιά. Θα να απαντήσω στους συναδέλφους και φίλους από την Παλαιστινή και τη Συρία. Ίσως υπάρχει κάποια παρεξήγηση, ίσως εγώ εκφράστηκα λάθος, μάλλον εγώ θα φταίω. Στόχος δεν ήταν το ψήφισμα. Το ψήφισμα ακολουθεί. Αργότερα θα έρθει το ψήφισμα. Στόχος μας ήταν να μην αφήσουμε να περάσει αυτή η συνεδρίαση σε καθεστώς σιωπής, δηλαδή να μην συζητηθεί καθόλου. Και είχα την εντύπωση σήμερα και από την πλειονότητα των παρεμβάσεων. Και ο κύριο Τολάμαν ήταν ε, απόλυτα σύμφωνα μαζί μου. Απόλυτα σύμφωνο μαζί μου. Και είπε προ το τέλο τη παρέμβασή του ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε προ ένα διάλογο. Έκανε έκκληση για διάλογο κτλ. Να κάνουμε έκκληση. για διάλογο. Ναι, αυτό είναι δηλαδή έκκληση για επανάληψη του διαλόγου έτσι ώστε οι κυβερνήσει να εισακούσουν του βουλευτέ. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το νόημα, όχι να επανέλθουμε. Όλοι τα γνωρίζουν όλα αυτά. Όλοι γνωρίζουν ε, τι ε, επιθέσεις έχουν υποστεί οι τι είδους ζημιές έχουν προκληθεί. Αυτό λέμε. Σημειώνουμε μόνο ότι συνεδριάσαμε, συζητήσαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης επευθύνθηκε αυτή η έκκληση. Και αυτό εν αναμονή του ψηφίσματος. Το ψήφισμα θα έχει όλες τις λεπτομέρειες, τα θέματα, τα σημεία κτλ. Και θα ικανοποιήσει όλες τις πλευρές, ελπίζω. Αυτό ήταν όλο. Τίποτε περισσότερο. Αν έπρεπε να συμπληρώσουμε το κείμενο με τέτοια σημεία, ήταν σαφέ ότι θα χρειαζόμασταν δύο ώρε συνεδρίαση παραπάνω. Και η πρόεδρο μου είπε ε, που δεν είδε να προλάβουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο γι' αυτό. Και περιοριζόμαστε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι θα διαφωνήσουν. Για την ελευθερία τη έκφραση και την ελευθερία τη θρησκευτική συνείδηση θα συμφωνήσω μαζί σας απολύτω και υπενθυμίζω τα λόγια της Ρόζας Λούξεμβουργκ. Ότι η ελευθερία δεν υπάρχει για κανέναν εάν δεν υπάρχει ελευθερία για αυτόν που έχει διαφορετική γνώμη. Αυτά. Και κατά τα άλλα συμφωνούμε. Άλλες παρεμβάσεις υπάρχουν, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και πάλι τους εισηγητές. Έκαναν εξαίρετο η δουλειά ως προς τη μέθοδο. Και το δεύτερο θέμα, οι τρεις εισηγητές έκαναν τη δουλειά, συμβιβαστική δουλειά, αν μπορώ να το πω έτσι. Έχετε ένα κείμενο στη θέσή σας. Σας παρακαλώ να το κοιτάξετε, να το εμπλουτίσετε. Αντιδράστε όπως θεωρείτε σκόπιμα. Σε συμφωνία με το άλλο θέμα, με τους, με τους ε, εισηγητές θα ετοιμάσουμε ένα κείμενο συμβιβαστικό κείμενο συμβασμού θα σας αποστείλουμε εγκαίρως πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Να το διαβάσετε λοιπόν εγκαίρως, να το εξετάσουμε στις 28 Ιανουαρίου στην προσοχή μας συνεδρίαση και εφόσον συμφωνείτε και αν έχουμε προχωρήσει αρκετά μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτές τις συμβαστικές θέσεις στην προσοχή συνεδρίαση. Πρόκειται και κείμενα τα οποία θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Εάν συμφωνείτε, Μπορώ να κηρύξω το πέρα τη συνεδρίασεως. Χαίρετε. Une qui s'est retournée.